Meine Damen und Herren, μου και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την συνεδρίαση. Υπάρχουν αλλαγές στην ενέργεια διάταξη, από ό,τι φαίνεται όχι. Οπότε καλωσορίζω εδώ πέρα τους βουλευτές που έχουν έρθει από την Αρμενία έχουν έρθει σε μια επίσκεψη λοιπόν. Καλώ ήρθατε. Περνάμε στο σημείο 2 και εκεί πέρα δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Και περνάμε στο σημαντικό σημείο το υπαριθμό 3 ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΕ κύριο Λαμπέρτο Ζανί. Πρέπει να πούμε πως ε, ήδη στην αρχή της θητείας σας είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας. Συζητήσαμε σημαντικά πράγματα για τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΑΣΕ και θέλω να ακούσουμε από σας τι γίνεται και τις ευρύτερες εξελίξεις από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαβιβοστόκ. Θεωρώ πως ακριβώς ε, μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη δραστηριοποίησή σας στον περιοχή Αφγανιστάν, Μογγολίας κτλ. Εκεί πέρα φαίνεται νομίζω ξεκάθαρα η ελκυστικότητα και η σημασία του ΟΑΣΕ. Βεβαίω, Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και μπρο. Έχουμε τη συνεργασία π.χ. στις ε, παρατηρήσεις εκλογών, στην κοινοβουλευτική διάσκεψη, τελευταία φορά στην Ουκρανία είχε συμβεί και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε αυτά. Να υπενθυμίσω πως πριν από χρόνια ναι, Είχαμε συνεργασία μεταξύ της κοινοβουλευτικής διάσκεψης του ΑΣΕ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούσε την ανάπτυξη της δημοκρατίας στα Βαλκάνια. Και τίθεται ερώτημα αν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε ξανά μια κοινή πρωτοβουλία για να κινηθούμε από κοινού σε κάποιες χώρες. Τώρα θα αλλάξει προεδρία από την Ιρλανδία, θα την, αναβάλει, ή θα την αναλάβει με η Ουκρανία. Και αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να αναλάβει την Προεδρία μια χώρα η οποία σύμφωνα με τα όσα είπαν οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ δεν εκπληρώνει τις, ε, τους όρους του ΟΑΣΕ για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά. Εδώ πέρα μας ενδιαφέρει λοιπόν η απόψη σας. Η συνεδρίασή μας είναι κοινή με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας ε, και Άμυνας αλλά και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οπότε θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στην κυρία Μπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Υποεπιτροπή μας ασχολούμαστε με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ένωσης και υπάρχουν πολλές χώρες εκεί πέρα που είναι μέλη του ΟΣΕ θα έλεγα. Πώς είναι, είναι κρίμα πως είναι διαρκές θέμα οι περιορισμοί των ΜΜΕ, αστυνομική κτηνοδία και, και σε χώρες εντό τη Ένωση υπάρχει διάκριση εις βάρος των Ρωμά και των Σύντη των μεγαλύτερων μειονοτήτων δηλαδή και εδώ πέρα φαίνεται πως η κατάσταση επιδεινώνεται. οπότε έχουμε μια χώρα η οποία δεν αφορά, μια κατάσταση η οποία δεν αφορά μόνο μια χώρα αλλά γενικώ. Οπότε εσείς στον ΑΣΕ έχετε κάποια φόρα συζητήσεων ε, που σας απασχολεί η κατάσταση των Ρωμά, το δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία, στη στέγη, αλλά και της μετανάστευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχαμε τη στρατηγική ενσωμάτωση των Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε πως ε, και από διεθνείς φορείς πρέπει να ασκηθεί πίεση για να πάρουν τα κράτη στα σοβαρά αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας uh, απευθύνω και πάλι το λόγο. Πριν από ένα χρόνο ήμουν μαζί σας ε, στο Στρασβούργο και αυτή η νέα ενημέρωση γίνεται την παραμονή της Υπουργικής ε, Συνεδρίασης ε, του Συμβουλίου που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία, διοργανωμένη από την ε, Ιρλανδική Προεδρία του ΟΑΣΕ. Στην ημερήσια διάταξη αυτής της Υπουργικής Συνέλευσης θα έχουμε διάφορες σημαντικές αποφάσεις. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο πακέτο αποφάσεων που αγγίζουν τα θέματα ασφαλείας όπως νέα μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, μια συζήτηση για την κυβερνοασφάλεια. Ξεκίνησε πριν από κάποιο χρόνο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα σε αυτή την διπουργική, αλλά πρόκειται για ένα διάλογο που εξελίσσεται καλά ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη και σίγουρα είναι και ένα θέμα που είναι σημαντικό για όλα τα κράτη ε, αν και βέβαια οι ε, προσεγγίσεις διαφέρουν, ωστόσο η συζήτηση αυτή βρίσκεται στο προσκήνιο διεθνώς και προσπαθούμε να βρούμε πιθανές συνεργασίες σε αυτό το τομέα. Έχουμε αποφάσεις στον οικονομικό επίπεδο αλλά και στο ανθρώπινο επίπεδο που αφορά το, ας πούμε, την ελευθερία των ΜΜΕ, το θέμα της ελευθερίας πρόσβασης στο ίντερνετ Επίσης μας απασχολεί ένα λεπτό ζήτημα για το οποίο υπάρχει αρκετά έντονη συζήτηση. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την ανοχή και την μη διάκριση. Πολύ σημαντικό θέμα θα έλεγα σε καιρούς όπου οι κοινωνίες συχνά ε, βρίσκονται διχασμένες, είναι διχασμένες για θέματα τέτοιου τύπου. Και υπάρχει και πάλι ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του Υπουργική Συνεδρίας που έχει να κάνει με την ευρύτερη και πιο μακρό πρόθεσμη συζήτηση που αφορά το μελλοντικό όραμα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια γενικότερα, από το πώς δηλαδή ε, σχετιζόμαστε Ποιε είναι οι απόψει των ΜΕΝ και των ΔΕ στο πλαίσιο αυτό το οποίο ορίστηκε από την διάσκεψη κορυφή στην ε, Στάνα πριν από δύο χρόνια ως ε, κοινότητα ε, ευρωατλαντικής και ευρωασιατικής ασφάλειας. Ποια δηλαδή είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή, πραγματικότητα, αυτή η πρόταση, αυτό το όραμα. Και ο διάλογος στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος ήταν τμήμα αυτής της διαδικασίας και θα συνεχίσουμε με πιο λειτουργικό τρόπο, ελπίζουμε μέσα στα επόμενα χρόνια, όπου στόχος θα είναι να έχουμε ένα σημαντικό σύνολο αποφάσεων, ε, τώρα το, ένα, κάποιο έγγραφο του οποίου μορφή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, για το 2015, όπου θα συμπέσει με την τελική πράξη του Ελσίνκη και την επέτειο αυτής θα συνδέσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή σε ένα θέμα της ημερησίας διάταξης στο Δουβλίνο και θα αρχίσει να δουλεύει η, επ' αυτού η ομάδα εργασίας. Ε, άλλη μια σημαντική απόφαση είναι βέβαια αυτή που ελήφθη μόλις την περασμένη εβδομάδα για την επέκταση μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερότητας να επεκταθεί ο οργανισμός αυτό μας ώστε να συμπεριλάβει και μια νέα χώρα τη Μογγολία η οποία μπήκε στην ΟΑΣΕ πρόσφατα και επισήμως θα προσχωρήσει στο Δουβλίνο. Αυξάνεται, μεγαλώνει λοιπόν η ΟΑΣΕ και το γεγονός ότι η Μογγολία προσχωρεί σε αυτήν θα τονίσει ακόμη περισσότερο ένα, μια πτυχή που είναι η ευρωασιατική πτυχή, η ευρωασιατική η ε, οπτική της ευρωπαϊκής ασφάλειας και βέβαια η συζήτηση και ο ρόλος που θα παίξουμε μέσω των αποστολών μας στην Κεντρική Ασία στην αντιμετώπιση του θέματος του Αφγανιστάν θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ΟΑΣΕ. Απλά και μόνο από οικονομικής άποψης να σας πω ότι η συμβολή των ευρωπαϊκών κρατών ανέρχεται στο 70% του συνόλου του προϋπολογισμού της ΟΑΣΕ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παίκτης κλειδί για την ε, ΟΑΣΕ. Και όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από την άποψη της θέσπισης πολιτικών και προτεραιοτήτων. Επίσης, εγώ δίνω μεγάλη σημασία στη σημερινή επαφή μαζί σας, γιατί έχω καταστήσει προτεραιότητά μου τη συνεργασία με τους ευρωβουλευτές, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, βέβαια που έχουμε κοινοβουλευτική συνέλευση. Έχω δει από την εμπειρία μου πόσο σημαντική είναι η κοινοβουλευτική διπλωματία εντό εισαγωγικών, δηλαδή να χρησιμοποιούμε οδούς, διάβλους διαφορετικούς από αυτούς που ε, είναι η παραδοσιακή κυβερνητική, ώστε να στηρίξουμε τους θεσμούς μας, να, έχουμε, να πετύχουμε μεγαλύτερη συνένεση, ε, να έχουμε επιπλέον δηλαδή συνεργασία που θα μας βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε πολύ συχνά δύσκολα θέματα. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και όλα σε αυτή την ευκαιρία, ώστε να δούμε λίγο και την ε, ημερήσια διάταξη του οργανισμού μας, καθώς προχωρούμε προς την Υπουργική... Ε, αλλά ε, να σας πω και πού υπάρχει σημαντική ευρωπαϊκή πτυχή. Να σας πω δηλαδή κάπως ποια είναι η εκτίμησή μου. Και αυτό με βάση το γεωγραφικό χώρο που λειτουργούμε, αν και καταβάλουμε πολύ ισχυρέ προσπάθειες ώστε να λειτουργούμε όσο γίνεται πιο οριζόντια και να αποφύγουμε τις διαχωριστικές γραμμές την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών ε, ε, σύμφωνα με γεωγραφικές περιοχές, αν δούμε την ε, πολιτική μας σφαιρικά, όπως ας πούμε στην πολιτική για τους ε, Ρώμα προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα και οριζόντια με σεβασμό για κάθε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη. Όπως σας είπα, θα ήθελα αυτό να το δομήσουμε, να δούμε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε επί τόπου. Νότια Ανατολική Ευρώπη είναι ο βασικός τομής, Δυτικά Βαλκάνια κυρίως, όπου επενδύεται το μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων μας επιτόπου. Στα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούμε να έχουμε τις μεγαλύτερες μας επιχειρήσεις. Το Κωσυφοπέδιο είναι το μεγαλύτερο με πάνω από 600 ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Αμέσως μετά ακολουθεί η αποστολή μας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Στην Νοτιοανατολική Ευρώπη εν γέννη θα έλεγα Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε δεσμευθεί επί τη βάση της εντολής που έχουμε Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα πιο δύσκολα θέματα. Η ευρωπαϊκή προοπτική εδώ είναι πολύ σημαντική λοιπόν, γιατί μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις μας λένε ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Οι προσδοκίες τους για ένταξη στην, ε, στα ευρωπαϊκά ή ευρωατλαντικά θεσμικά όργανα και μας ζητούν να περιλάβουμε εκεί στάνταρ τα οποία θα τους βοηθήσουν να προσχωρήσουν στους οργανισμούς αυτούς ε, πιο γρήγορα. Ενώ δηλαδή προσπαθούν να αναπτυχθούν, προσπαθούν να δουν, προσπαθούμε να δούμε το ρόλο μας ε, όχι για να βοηθήσουμε κάθε μια χώρα, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε Βοηθάει αυτό και γι' αυτό το λόγο και έρχομαι συχνά στις Βρυξέλλες, συζητώ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την Κομισιόν κάθε φορά και μαζί σας φυσικά, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όχι μόνο υπάρχει καλή συνεργασία, αλλά και στρατηγική σύγκληση. να συζητήσουμε ποια είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουμε τους πόρους που επενδύουμε επί τόπου. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτό τον καιρό χαλεπό, το χαλεπό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις και να επενδύουμε χρήματα στους τομείς όπου ε, είναι αναγνωρισμένες οι προτεραιότητες. Να αναφέρω σύντομα λοιπόν κάποια από τα θέματα. Πρόσφατα επισκέφθηκα την Αλβανία και είχα εκεί επαφές με τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση. Ήταν μια ευκαιρία για μια πραγματική ε, συνάντηση με την κυβέρνηση παρατήρησα πραγματική πρόοδο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Έχουν γίνει πραγματικές προσπάθειες, έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες που θα οθήσουν την Αλβανία πιο κοντά, να έρθει πιο κοντά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης καταγράψαμε τι πρέπει ακόμα να γίνει δουλειά για μεταρρυθμίσεις, δουλειά για πλήρη εμπλοκή και δέσμευση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και του Κοινοβουλίου, εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει πρόσφατα περάσει. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας, Ανησυχήσαμε για κάποιες από τις πρόσφατες εξελίξεις επιτόπου γιατί υπάρχουν ε, σημεία σημάδια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις κοινότητες ε, έχουν γίνει πιο περίπλοκες και πιο τεταμένες. Ε, ε, γι' αυτό πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει η χώρα αυτή. Εμείς από την δική μας πλευρά συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά επιτόπου. Βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό στα Σκόπια αλλά ίδια κάποια παρόμοια δυναμική και στη Βοσνία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε επιτυχίες στις διεθνείς, στις διεθνούς ο Οχρίδα και Ντέιτον. Επιτυχία στο να σταματήσει η σύγκρουση και να επιβληθεί σταθερότητα. Αλλά Υπήρχαν κάποια πλαίσια που προστάτευαν τις ε, μειονότητες και τις ε, εθνοτικές μειονότητες αυτές τις χώρες. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς που έχει βασιστεί σε αυτά τα εργαλεία, διαπιστώνουμε ότι η παρατεταμένη εφαρμογή αυτών των συμφωνιών στην ουσία παράγει μεγαλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα στις κοινότητες. Είναι δηλαδή πια ο καιρός να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιβληθούμε ε, πάνω από αυτά ε, τα στοιχεία, να βρούμε δηλαδή νέα στοιχεία που θα φέρουν κοντά τις δύο κοινότητες και θα κάνουν τις χώρες αυτές πιο βιώσιμες ε, και τις σχέσεις ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες πληρέστερες και πιο παραγωγικές. Στο Κωσυφοπέδιο, όπως ανέφερα, έχουμε ακόμα τη μεγαλύτερη συνεργασία. Στηρίζουμε απόλυτα τον διάλογο που έχει ξεκινήσει από την... και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε πως οι ευρωπαϊκές προοπτικές είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο που θα διευκολύνει την ε, πρόοδο για την αντιμετώπιση δηλαδή των θεμάτων που ανακύπτουν οι ΟΑΣΕ, δεσμευμένοι τόπου Έχουμε ισχυρέ σχέσεις με τις κοινότητες. Είμαστε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε και συμφωνίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει μέσα στην πλαίση, στο πλαίσιο του διαλόγου να διευκολύνουμε τις επαφές ανάμεσα στις... Ε, μάλλον έχουμε μάλλον διευκολύνει τις σερβικές κοινοβουλευτικές εκλογές στο Βόρειο Κόσοβο, το οποίο έχει στηριχθεί και από τη σερβική πλευρά και από την πλευρά του Κωσυφοπεδίου. Ε, εξετάζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και βλέπουμε και πού μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Η Σερβία έχει την προεδρία, θα έχει την προεδρία μάλλον το 2015 που θα είναι η του, 14η επέτειος του Ελσίνκη. Η Σερβία θα έχει τότε και την προεδρία της ΟΑΣΕ και άρα και το έργο του να καταλήξει σε συμπεράσματα αυτή η διαδικασία του μέλλοντος της ε, ο ΑΣΕ από τώρα είναι πολύ δραστήριο μέλος ε, της κοινότητας χωρών της ε, ΟΑΣΕ και ακόμα εμείς δουλεύουμε στην ε, στο Βελιγράδι και προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καλή μας συνεργασία. Η Βοσνία παραμένει περίπλοκη. Ε, δεν έχουμε δει πολύ πρόοδο πρόσφατα. Δεν είναι εύκολο να εμπλακεί και να συνεργαστεί η διεθνής κοινότητα και αυτό οδηγεί σε απόγνωση γιατί οι πρόοδοι που θέλαμε να σημειωθούν λείπουν ακόμη. Διάφορες πρωτοβουλίες ε, όπως η αντιμετώπιση ε, του, των προβλημάτων είναι δύσκολη γιατί δεν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες ακόμα και όταν περνούν. Είναι ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε, προσπαθούμε, επιμένουμε. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται δεν εφαρμόζονται στο τέλος. Ε, πάντως επιμένουμε, επιμένουμε ε, και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με ε, την χώρα. Τώρα, πιο ανατολικά στη Μολδαβία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στη διαδικασία 3 συν 2. 5 συν 2, με συγχωρείτε. Μαζί με τη Ρωσία και την Ουκρανία η οποία η Ουκρανία θα έχει την Προεδρία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος. Έχουμε την Προεδρία της ΟΑΣΕ του χρόνου. Και ως βασικός παίχτης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις αναμένουμε η Ουκρανία να εμπλακεί πλήρω στη συνέχιση αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία 5 συν 2 ξεκίνησε το περασμένο χρόνο μετά από μια διακοπή 5 ετών περίπου. Ξεκίνησαν καλά, κινήθηκαν γρήγορα, νέα ηγεσία ήταν δεσμευμένη και ε, προσιλωμένη και έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου τώρα πιο δύσκολα θέματα έρχονται στην ημερήσια διάταξη και αυτό συμπίπτει τις τελευταίες μέρες με κάποια οπισθοχώρηση ή μάλλον μια επιβράδυνση της διαδικασίας. Όπως σας είπα, καθώς στάσαμε σε κάποια λεπτά ζητήματα, χρειάζονται σταθερές και επίμονες προσπάθειες και είναι ένας τομέας όπου η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχιστεί με πολύ συντονισμένο τρόπο. Λευκορωσία. Στην Λευκορωσία αναπτύσσεται ένα πακέτο Έχουμε κλείσει την αντιπροσωπεία μας στο Μίνσκα πριν από δύο χρόνια, λίγο παραπάνω από δύο χρόνια. Και δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Εκτότε φυσικά η Λευκορωσία είναι προβληματική από πολλές απόψεις και για μας. Οι δικές μου σχέσεις με την ηγεσία είναι τελείως επιφανειακές και ε, πολύ ε, πρόσχερες, αλλά Έχουμε κάνει ένα σχέδιο δραστηριότητας που καλύπτει όλες τις διαστάσεις συμπεριλαμβανομένες τη ανθρώπινης και αυτό το έχουμε καταστήσει ως όρο. Μόλις το δέχτηκε η αντίστοιχη προσωπία της Λευκορωσίας, δεν βλέπουμε ποια θα είναι οι δραστηριότητε αυτές για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε τις συνεργασίες. Σε ορισμένους τομείς προσπαθούμε να δούμε μέχρι πού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για παράδειγμα, έχουν ε, τις Εκλογές. Ε, παρακολουθήσαμε τις εκλογές, μόλις εξεδόθη δε μια ανέκθεση και αναμένουμε η κυβέρνηση Λευκορωσίας να συνεργαστεί για την εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Παρομοίως και με την Ουκρανία θα δούμε ποια θα είναι η τελική έκθεση, αλλά θα πρέπει να πω εν γέννη και τελικά ότι δεν θέλω να περιπλακεί το θέμα της Προεδρίας της Ουκρανίας, της ΟΑΣΕ, με τα θέματα της ίδιας Ουκρανίας ή των σχέσεων της Ουκρανίας με άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την Προεδρία και την προετοιμασία για την Προεδρία, με χαρά είδα πως η Ουκρανία είναι πολύ αφοσιωμένη και δεσμευμένη, κάνει καλή δουλειά. Οι διαβουλεύσεις με την Ουκρανική ηγεσία μέχρι στιγμής για την Προεδρία του ΟΑΣΕ είναι την επιτυχής. Η Ουκρανική πλευρά <clears throat> λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το θέμα και προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά. Ε, είναι εξοικειωμένη με τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη του οργανισμού μας και μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο. Φυσικά άκουσα τα όσα έλεγε ο πρόεδρος για το κατά πόσο η Ουκρανία ή μάλλον πού βρίσκεται η Ουκρανία όσον αφορά την εφαρμογή των δικών της δεσμεύσεων αλλά αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους συμμετέχοντες αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος κανόνας μέσα στην ΟΑΣΕ ώστε να παρεμποδίζονται χώρες επί τη βάση τη στήριξη των δεσμεύσεών του ή όχι. Ο ΣΕ είναι ένας ανοιχτός οργανισμός και κάθε χώρα έχει πρόσβαση στην Προεδρία και είναι ευπρόσδεκτη σε αυτήν να παίξει ρόλο. Αλλά σίγουρα με αυτόν τον τρόπο η κάθε χώρα δέχεται ότι θα λειτουργήσει ως μοντέλο, ως πρότυπο. Και αυτό θα είναι το ίδιο μια πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση της Ουκρανίας. Γεωργία και Νότιος Κάφκασος γενικότερα. Πολύ λίγες εξελίξεις. Οι διαπραγματεύσεις της Γενέβης δεν έχουν ε, βοηθήσει στην πρόοδο, ωστόσο έχει υπάρξει ειρηνική μετάβαση της εξουσίας μετά από μια πολύ έντονη και ε, εκστρατεία η οποία δίχασε τον κόσμο. Με περηφάνεια σας λέω ότι ήμασταν παρόντες, παρακολουθήσαμε, παίξαμε το ρόλο μας στην εξασφάλιση και ενός κλίματος ειρηνικής αλλαγής κυβέρνησης. Υπάρχουν ακόμα φυσικά προκλήσεις και μιλάμε με την κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα που εμείς διαπιστώνουμε, αλλά εν γέννη έχει εξελιχθεί η κατάσταση θετικά. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει προβληματικό. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτή τη στιγμή. Μετά από, από την υπόθεση Σαφάροφ στο Αζερβαϊτζάν, και τώρα γίνεται λόγος για άνοιγμα ενός αεροδρομίου στον Αγκόρνο Καραμπάχα που είναι επίσης δυνητικά προβληματική υπόθεση και θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις. Επί τόπου τέλος, Κεντρική Ασία έχουμε πέντε επιχειρήσεις στα πέντε κράτη, σε πέντε κράτη. Κεντρική Ασία, βασικό στρατηγικό στοιχείο είναι το γεγονό ότι εστιάζουμε του στο Αφγανιστάν ω αποτέλεσμα απόφαση που ελήφθη στην Υπουργική του Βίλνιου πέρυσι Εστιάζουμε λοιπόν στο Αφγανιστάν και την έμφαση για να αντιμετωπίσουμε το Αφγανιστάν κάπως όπως το πνεύμα της διαδικασίας της Ισταμπούλ, δηλαδή να βοηθήσουμε τα συμμετέχοντα κράτη της Κεντρικής Ασίας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από το Αφγανιστάν, από ωραίων από το Αφγανιστάν, ας πούμε, ασφάλεια των συνόρων, οι ρίζες ε, ε, αίτια όπως ας πούμε η παιδεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και θέματα σχετικά με την τρομοκρατία. Άλλο τρόπο λειτουργία είναι να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε να έχουν επαφές με το Αφγανιστάν και να παρεμβαίνουν για τη σταθεροποίηση της χώρας, ειδικά μετά από το 2014, όπου ο ρόλο της διεθνούς κοινότητας στο Αφγανιστάν θα αλλάξει. Δύο λόγια τέλος για τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, με τους ε, μεσογειακούς μας εταίρους σχέσεις του ΣΟΑΣΕ τελευταία είναι πιο επιχειρησιακή, πιο λειτουργική. Είναι περισσότερο, παλιότερα ήταν περισσότερο πολιτικός διάλογος, ενώ τώρα παίρνει μια μορφή ε, πιο επιχειρησιακή, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από αυτές τις χώρες και ε, ενδιαφέρονται για δικέ μας εμπειρίες, για τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει, για την πείρα μας όσον αφορά τη δημοκρατική μετάβαση και συζητάμε μαζί τους τώρα για προγράμματα δράσης, σχέδια δράσης που θα περιλαμβάνουν βοήθεια σε τομείς εμπειρογνωμοσύνης για παράδειγμα. Και για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών θεσμών ε, στην Βαρσοβία που υπάρχει σε υπηρεσία, οπότε τώρα θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε μια τελεία και είδατε επομένως κάναμε ε, έτσι μια σχεγράφηση των βασικών θεμάτων και θα συνεχίσουμε αν υποβάλλετε ε, τυχόν ερωτήσεις για ό,τι σας ενδιαφέρει. Ο πρώτος ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Πέτερλα. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, με μεγάλη μας χαρά Έχουμε τη σημερινή συζήτηση για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος ε, δίνει σημασία στο αποτέλεσμα και ε, εάν κάτσουμε και δούμε όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και βέβαια μας τα παρουσιάσατε με ένα σωρό μεταβλητές αισιόδοξε, τελικά όλα αυτά μας άγουν στο ε, ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα και να μπορέσουμε ο φορέας σας να έχει ουσία, να έχει αποτελέσματα και έτσι να σταθούμε επιτυχία οι προσπάθειες. Επομένως, ε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Βλέπετε να, να, να ξανοίγονται κάποιες ευκαιρίες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο στενή συνεργασία εμείς και εσείς και έτσι να έχουμε στη δουλειά μας προσθεμένη αξία. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ευκαιρίες που ξανοίγονται σε εκτελεστικό, κυβερνητικό ας το πούμε επίπεδο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ε, καταστάσεις, κάποια σημεία στα οποία έχουμε κολλήσει κατά τον τρόπο, όπως είπατε για την Μακεδονία λέω μιλτής, και ότι ε, είναι, είναι, είναι, είναι ορατό ε, είναι αισθητό το ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει ορισμένα σημεία και άρα θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιες πολιτικές και μάλλον αρνητικές πολιτικές συνέπειες που αναδύονται. Για πέστε μας επομένως, τι, ο οργανισμός σας, τι μπορεί να κάνει σε αυτή την λεγόμενη προληπτική διπλωματία, γιατί βεβαίως καθ' αυτόν τον τρόπο έχουμε ε, πολλές διαφορετικές επιλογές. Πάντως θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο μας ε, ενδιαφέρει πολύ, το οποίο το ε, αγαπάμε. Είναι ο κοινό μα έρωτα, είναι το, το, το Κυργιζιστάν. Για εκεί, τι λέτε, τι, θα χρειαστεί να κάνουμε παραπάνω. Και πάλι σα ευχαριστώ εκ των προτέρων και για τι απαντήσει σα. Επόμενο. Γκόμε. Σα ευχαριστούμε για την εισήγησή σα. Παρακαλώ, πέστε μας ε, λίγο λόγια παραπάνω από την κυβερνοασφάλεια. Ε, τι, τι κάνουν, ε, τι, τι κάνει ο οργανισμός σας, τι, τι, τι, πού, πού διαφέρουν οι απόψεις μας. Αν μπορείτε, πέστε μας δύο λόγια για το τι εξέλιξη έχουμε όσον αφορά την ελευθερία προσβασιμότητας, αλλά επίσης πώς θα μπορούσαμε αυτή την κυβερνοασφάλεια να τη χρησιμοποιήσουμε σαν όπλο. Ας πούμε το 2007 είχαμε την περίφημη κυβέρνηση επίθεση στην Εσθονία. και άρα πρέπει να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Τώρα, άλλο θέμα. Εμείς. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιε είναι οι συνέπειε τη λιτότητα. Ποιο είναι το κόστος τη λιτότητα όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός μας. οπότε για τα βασικά σα θέματα, τα δικά σα ή τα θεμελιώδει αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλώ γενικότερα πλευρά δημοκρατία. Το κόμμα το ναζιστικό που έχει μπει στο κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω και που επιτίθεται ει του μετανάστε και επομένω. Τι λέτε, τι, τι, τι λέει ο οργανισμό σα. Τέλος, δε. Για πέστε μας όσον αφορά την τόσο αισιόδοξη αποψή σας για την Ουκρανία και πέστε μας όσον αφορά την Λευκορωσία αλλά και την Ρωσία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Ε, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΑΣΕ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε ε, ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι άμεσα αιρετό. Συνεργαζόμαστε όμως ε, με τον ΟΑΣΕ σε αποστολές παρατήρησης εκλογών και εκεί πέρα δυστυχώς δεν είναι ιδανική η συνεργασία. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένω από το Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτική διάσκεψης του ΟΑΣΕ να έρθει εδώ για να δούμε τέτοιες συνεργασίες. Και θα σας παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε τους εσωτερικούς διάβλους του ΟΑΣΕ για να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι δεύτερον. Ότι βεβαίω η υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που είναι ιδιαίτερο σεβαστή και επαγγελματική στον τομέα της δημοκρατίας και της ε, αποστολής των εκλογών. Τα μιλάτε για τις χώρες εταίρους στη Μεσόγειο και κάποια πράγματα τα οποία γίνονται επιχειρησιακά, ε, μιλάτε και για εκλογές. Υπάρχει μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΟΑΣΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο ΑΣΕ δεν κάνει παρατηρήσεις εκτός της, της ε, περιοχής του και αντιστρόφως. Δυστυχώς στη Βόρεια Αφρική, ο ΑΣΕ έστειλε μια μεγάλη αποστολή στην Τινησία, κάτι το οποίο δημιούργησε σύγχυση. Γιατί όπως σας είπα δεν είναι και φοβερή η φήμη της κοινοβουλευτικής διάσκεψης του ΑΣΕ. Πρέπει λοιπόν ο ΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο υψηλότερο επίπεδο να επανα αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ήταν ιδιαίτερα σημαντικός εδώ και χρόνια και θα σας ενθάρρυνα να το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στη χώρα μου ε, υπάρχει, μεγάλη, υπάρχει μεγάλη αντίσταση στον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάρχουν ακόμα και ανοιχτές προτάσεις για να αποσυρθούμε από την ΕΣΔΑ. Αναρωτιέμαι πως υπάρχουν κάποιες σκέψεις ε, για να συμφωνηθεί ο ΑΣΕ με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, θα γλιτώναμε πάρα πολλά λεφτά έτσι και έτσι θα είχαμε μια περιοχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Βόρεια Αμερική μέχρι την Κεντρική Ασία. Σκέφτεστε κάτι τέτοιο. Κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Γενικό Γραμματέα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα. Τι ισχύει όσον αφορά την θέση της Ρωσίας. Όπως το γνωρίζουμε. Η συμπεριφορά και η στάση δεν συνάδει προς τις αρχές της οργανωσίας σας κύριε Γενικέ. Για μας, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, κάποια αλλαγή τα τελευταία χρόνια και προς τα πού πάει το πράγμα. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε, εάν ε, τώρα, τον τελευταίο καιρό, στην ε, υπηρεσία σας, έχετε προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή προς αυτή την εξέλιξη, κάτι το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και όλα τα μέλη του οργανισμού σας. Και πολλοί ακολουθούν μεροληπτική πολιτική, είτε πρόκειται περί κάποιου είδους ε, σιωπή όσον αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους ή όσον αφορά πάλι την αδράνεια, τη σιωπή, όσον αφορά τα τόσα ανησυχητικά που γίνονται στην Γεωργία. Για πέστε μου, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ. Το Καζακστάν το 2010 είχε την προεδρία του ΟΣΕ και είχε υποσχεθεί πως όλες οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα γίνονταν σεβαστές, αλλά μετά από την ε, Προεδρία η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώθηκε και πάλι. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε πως ε, ανεξάρτητα ΜΜΕ στο Καζακστάν εμποδίστηκαν. Πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν ε, για εσάς ε, έκανε το Καζακστάν αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια πράγματα για τα οποία είπατε για την κυβερνοασφάλεια και την ελευθερία στο διαδίκτυο και να σας ρωτήσω για το πώς ε, βλέπετε την ισορροπία και να μην υπάρχει βεβαίω ότι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος θεωρείτε πως υπάρχουν περισσότερες ε, ευκαιρίες για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ποιες είναι οι απειλές κατά την άποψή σας. Εγώ ήμουν κυρίω σε επαφή με την κυρία Μεγιάτοβιτ, εκπρόσωπο για την ελευθερία των ΜΜΕ και κάνει εξαιρετική δουλειά. Έθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπατε για την Ευρασία πώς βλέπετε την Τουρκία, μια χώρα με προκλήσεις όσον αφορά την ελευθερία ΜΜΕ, λόγου και διαδικτύου, αλλά και ευρύτερα. Φιλόδοξο παίκτη σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο της Τουρκίας και τρίτον, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η κυρία Νάιτς, θεωρώ πως όλοι προσπαθούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΣΕ με την έννοια της αρισιμότητας και των δεσμεύσεων που κάνουν τα κράτη-μέλη αλλά και το τι ε, έχουμε εμείς ως μοχλοποίηση εναντίον των άλλων. Ποιος είναι για σας ο αποτελεσματικότερος τρόπος έτσι ώστε τα μέλη αλλά και οι χώρες που σχετίζονται με τον ΟΑΣΕ να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οικονομική τους δύναμη για τις αξίες που συμμεριζόμαστε αλλά δεν τηρούνται πάντα ούτε καν από τα μέλη μας πόσο πάλι από τρίτες ε, χώρες. Ευχαριστώ. Και Γιάννης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια πρώτη σκέψη. Ότι τα όσα είπατε κύριε Γενικέ επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο εγώ πρεσβεύω εδώ και καιρό ότι δηλαδή οι πολυμερείς διπλωματία και οι μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη αλλά και πέραν της Ευρώπης μετά από τον ε, Μεγάλο Πόλεμο ε, χαρακτηρίζονται σαν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της ανθρωπότητας για τον 20ο αιώνα. Και αυτό επίσης ε, αποδεικνύεται και στο Συμβουλίο της Ευρώπης, αυτό που είναι και από τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του οργανισμού σας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η στόχη σας ε, και βεβαίω, όπως και εγώ και άλλοι υπερασπιζόμαστε τον οργανισμό γιατί επιτελεί τέτοιο έργο. Και κάποιος ε, συνάδελφο κάτι είπε, επέκρινε τέλο πάντων το Συμβουλίο τη Ευρώπη, αλλά δεν συμφωνούμε όλοι με αυτά, με του τα επικριτικά λόγια. Και βεβαίως ε, κατά μείζον λόγω αυτά ισχύουν και για τον φάρο ελευθερίας, αξιών, ελευθεριών που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βεβαίως ε, αποτελεί το τον προμαχώνα για να υπερασπιστεί κανείς τα δικαιώματά του και έναντι του κράτους. Επομένως, δεν θα πρέπει με διάφορους τρόπους να υπονομεύουμε το έργο των αυτών των θεσμών. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα ΜΜΕ, ε, τι γίνεται ας πούμε με τον Βρετανικό τύπο, γιατί μιλώ μόνο για τα ταμπλόιτς. Ε, έχει γίνει μια διολίσθηση προς τον ε, λαϊκισμό και αυτό αφορά επίσης όχι μόνο καν την Βρετανία. Έχουμε κάποιες ε, αντιδραστικές δυνάμεις που ακριβώς συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο να υπονομεύουν δηλαδή αυτούς τους δεσμούς και εκτός Βρετανίας. Τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καθώς έχετε αρκετή εμπειρία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το ζήτημα των συνοριακών ζητημάτων ως ένα ζήτημα που πρέπει να επιληθεί κατά προτεραιότητα στην διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης. Πράγματι υπάρχουν αρκετά άλλη τα προβλήματα και βεβαίω είναι πολύ συναισθηματικό ζήτημα. Προσφάτως είχαμε την απόφαση του δικαστήριου της Χάγης και αναρωτιέμαι εάν ο ο ΑΣΕ μπορεί να δράσει προληπτικά σε ζητήματα συνοριακά μεταξύ των χωρών της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Ευχαριστώ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να, να τις απαντήσω. ξεκινώντας από τον κύριο Πέτρελε για το πώς θα αποκτήσει περισσότερη δύναμη ο ΑΣΕ. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε βεβαίως, αφενός συζητάμε εντό του ΑΣΕ και έχουμε και αποφασίσει για την ενδυνάμωση του οργανισμού, οπότε και εμείς Βεβαίω ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας, αλλά βεβαίως η ουσία είναι τα κράτη-μέλη τα οποία κάποια στιγμή θέτουν κάποια όρια. δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από αυτά τα οποία θέλουν τα αφεντικά μας. Αν δείτε παραδείγματος χάρη την προληπτική διπλωματία. Στην προληπτική διπλωματία αυτό το οποίο θα έλεγα είναι πως δώστε μας ένα ρόλο στην αρχή μιας κρίσης ε, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Π.χ. να κάνουμε κάποιες ε, συστάσεις ε, για να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο. Βεβαίως το ζήτημα είναι πως όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν υπάρχει μια καλή προεδρία και η Προεδρία έχει συνένεση. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μία φορά, αλλά εάν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο θεσμοποιημένο σε μόνιμη βάση ε, δεν θα τα καταφέρουμε και αυτό το συζήτησα και με τον ε, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Μπαν Κιμούν που το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει κανεί δεν δίνει επιταγή εν λευκό σε έναν διεθνή οργανισμό για να κάνει αυτό το οποίο λέμε προληπτική δράση υπάρχει μια λεπτή, ευαίσθητη ε, γραμμή μεταξύ έγκαιρης προειδοποίησης και έγκαιρης δράσης. Η έγκαιρη δράση πρέπει να εγκριθεί από τις χώρες, οπότε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και κάθε φορά πρέπει να δούμε τι πολιτικό περιθώριο έχουμε. Μία επιλογή είναι βεβαίως οι ε, συνεργασίες. Ε, τώρα στην Κυργυζία εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες ανησυχίες, ειδικά στο Νότο. Εξακολουθούμε να έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση που εστιάζεται στην πολυεθνική αντιπολίτευση της περιοχής και να μην υπάρχει διάκριση από την αστυνομία, λέγεται η πρωτοβουλία ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στηρίζει και σκέφτεται βέβαια περαιτέρω στήριξη και με της ευκαιρίας να σας ενημερώσω γι' αυτό για να υπάρξει και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δουλειά που κάνει ο ΑΣΕ τις πολύ αυτές τις περιοχές. Κυβερνό ασφάλεια. και τα σχετικά ερωτήματα. Υπάρχει εδώ πέρα μια συζήτηση για το που είναι το όριο. Και είναι δύσκολο ζήτημα, αν και βεβαίως δεν εμφανίζεται τα στα έγγραφα τα οποία μας ασχολούν. Και το ζήτημα είναι περισσότερη ασφάλεια ή περισσότερο άνοιγμα και πρόσβαση, ελευθερία πρόσβασης. Και η συζήτηση ξεκινάει ήδη από την ορολογία και τους ορισμούς το πώς ορίζεται η ασφάλεια του διαδικτύου. Η προσέγγιση που έχουμε στον ΑΣΕ είναι σχετικά ήπια. Εξετάζουμε την ασφάλεια ως ε, το νέο σύνορο της ασφάλειας των κρατών μελών και έχουμε την λεγόμενη ήπια ασφάλεια όπως λέγεται για να αναπτύξουμε κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, π.χ. άμεση πληροφόρηση, ε, όταν υπάρχει επίθεση, διαβεβαιώσεις και κάποια άλλα ζητήματα που είναι πολύ τεχνικά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως ε, η ελευθερία των ε, ΜΜΕ σημαίνει πως θα παρακολουθούμε αυτή την συζήτηση και οπωσδήποτε πολλά κράτη-μέλη και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι μέρος αυτής της συζήτησης είναι ενεργοποιημένα και παρακολουθούν που πάει αυτή η συζήτηση. Για το θέμα τώρα του τι σημαίνει η λιτότητα και τα αποτελέσματά της θεμελιώδεις αξίες ε, και την ε, δημοκρατία. Κοιτάξτε, ο ΑΣΕ πρώτα απ' όλα είναι ένας οργανισμός ασφαλείας. Η προσέγγισή μας βασίζεται στην ανάγκη να ενισχύσουμε την ασφάλεια στο χώρο του ΑΣΕ. Αλλά αυτό γίνεται επί τη βάση μιας ευρύτερης προσέγγισης που βεβαίως συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αλλά και την οικονομική ανάπτυξη και τα, και τα ζητήματα ασφαλείας βεβαίως. Το ζήτημα λοιπόν των θεμελιωδών αξιών και το πώς ε, εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη. Ο ο ίδιος ε, δίνει τη δυνατότητα όλων σε τον χρόνο της χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τους δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουν το πώς άλλα κράτη-μέλη του οργανισμού ε, αντιμετωπίζουν την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους. Και είναι πολύ έντονος ο διάλογος, συνεχής και καμιά φορά και αρκετά έντονος με πολλές διαφωνίες. Αλλά αυτό είναι κάτι το υγιές, γιατί πράγματι κάπου εκεί μπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση σε βάση εβδομαδιαία ή ακόμα και ημερήσια. Οπότε ο ΑΣΕ είναι ένα μέρος που αξιολογούμε ο ένας τον άλλον και υπάρχουν διαφορετικές αξιολογήσεις βεβαίως. Και υπάρχουν και κάποιες πολύ, πολύ έντονες ε, συζητήσεις. Υπάρχει αίσθηση ως κάποιες χώρες ε, οπισθοχωρούν. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες χώρες ε, που περιμένουν ε, από τη μία μέρα στην άλλη δημοκρατικό μετασχηματισμό σε κοινωνίες όπου χρειάζεται μια αλλαγή γενεάς για να βελτιωθούν τα πράγματα. Και σημασία έχει η κατεύθυνση, αλλά καμιά φορά και η κατεύθυνση δεν υπάρχει. Οπότε εκεί πέρα είναι πιο προβληματικά τα πράγματα. Αλλά για να επανέλθω στην λιτότητα. Εμείς είμαστε ένας φτηνός οργανισμός, έχουμε έναν προεκλογισμό 140 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε 16 επιχειρήσεις. Οπότε οπωσδήποτε δεν ε, είμαστε από τους οργανισμούς που κοστίζουν. Αν δείτε συνεισφορές ε, Συχνά ε, είναι, ο προπολογισμό μας δηλαδή είναι αυτός μίας ειρηνευτική αποστολή. η κοινοβουλευτική διάσκεψη. Έχουμε και εσωτερικά προβλήματα, ειδικά προσφάτως με τις εκλογές στις ΗΠΑ όσον αφορά την, ε, την υπηρεσία δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Η κοινοβουλευτική διάσκεψη είναι κάτι το αυτόνομο και η φύση της ακόμα είναι κάτι συζητήσιμο. Υπάρχουν απόψεις για το τι ακριβώς είναι και πώς σχετίζεται με τις δομές αυτές. Αλλά δεν είναι μία από τις δομές του ΩΣΑ και κατά κάποιον τρόπο εωρείται, αν θέλετε, η φύση του, του Εγώ θέλω, όπως είπα, μια δυνατή ισχυρότερη σχέση μεταξύ ημών και ημών. Το ζήτημα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς προέκυψε. Εγώ δεν θα έλεγα πως είναι πολιτική του ΟΑΣΕ, αλλά οπωσδήποτε περιλαμβάνει την υπηρεσία δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ε, οπωσδήποτε θα το θέσω με τον διευθυντή της υπηρεσίας, αλλά εγώ δεν έχω δει το γραφείο αυτό να κάνει κάποιες ε, πράξεις ή να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, γιατί... Ε, μην ξεχνάτε πως, ε, όπως είπα, η κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΟΑΣΕ είναι κάπως αυτόνομη. Οπότε το είδα αυτό, είδα την έκθεση και τα λοιπά, αλλά ε, ήταν, ήταν η κοινοβουλευτική διάσκεψη. Αυτό το οποίο κάνει η Υπηρεσία Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων είναι να απαντά σε αιτήματα βοήθειας, π.χ. πώς δίνονται ε, εκλογικές επιτροπές ε, λοιπά. Ε, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως πάμε σε αποστολές παρατηρήσεις εκλογών. Είναι κάποια βοήθεια και είναι κάποια από τις βοήθειες για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και πάλι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ταυτίζεται ε, με τον ΟΑΣΕ, γιατί εμείς είμαστε οργανισμός ασφαλείας, ε, ασχολούμαστε με έλεγχο όπλων κτλ. Το ΟΔΙΡ όμως, η υπηρεσία όπω είπα ανθρωπινών δικαιωμάτων και δημοκρατία. Ε, ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Έχουμε και τον απεσταλμένο για την ελευθερία των ΜΜΕ. Οπότε το εξετάζουμε για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και συνέργεια. Και αυτά κάνουμε. Δεν υπάρχει εξετάζουμε τη συγχώνευση, το Συμβούλιο της Ευρώπης έκανε μία μελέτη για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Εάν ε, πρέπει να γίνει κάτι δραστικότερο, αυτό νομίζω επαφίεται στα κράτη-μέλη των διοργανισμών. Πρέπει να έχετε κατά νου πως ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Έχουμε κάποιον διευρωπαϊκό δεσμό, διατλαντικό δεσμό, δηλαδή τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Και βεβαίω ε, και μια σχετική διάσταση τώρα που έχει ενταχθεί και η Μογγολία. Για τη Ρωσία σας παραπέμπω σε αυτό το οποίο είπα. Εγώ δεν θέλω να κάνω αξιολογήσεις, αλλά βλέπω τις συζητήσεις και υπάρχουν συζητήσει, όπω είπα για την αντιμετώπιση των ΜΚΟ, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία του συνέρχεστε κτλ. Οπότε παρακολουθώ αυτές τις συζητήσεις. Και βεβαίω. Βλέπουμε και επιλεκτική χρήση της δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν κάνουμε διαβουλεύσεις με χώρες όπου βλέπουμε τέτοιες απόπειρες, πάντα παρεμβαίνουμε και μιλάμε σε εκπροσώπους της κυβέρνησης και επισημαίνουμε ξεκάθαρα πως δεν είναι αποτεκτές αυτές οι πρακτικές. Για το Καζακστάν Όπως είπα, δεν κρίνουμε μια χώρα πριν ε, τη δεχτούμε ε, και την αναλάβει την Προεδρία. Θα έλεγα πως ε, εκ πως ήταν θετικό το να έχει το Καζακστάν την Προεδρία. Ε, κατέβαλαν λοιπόν μία προσπάθεια και ενεργοποιήθηκαν εντός ε, του οργανισμού όλοι, όλα τα θέματα της Κεντρικής Ασίας απασχόλησαν πολύ περισσότερο τον οργανισμό Είναι λοιπόν περιπλοκή κατάσταση. Όπως σας είπα, πράγματα καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και χρόνος, γιατί μιλάμε για κοινωνίες πολύ διαφορετικές, που έχουν τη δική τους ιστορία και όπου η αλλαγή θα απαιτήσει χρόνο. Δεν, δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια εύκολη λύση. Χρειάζεται απλά μία στήριξη μόνιμη, μια εμπλοκή μόνιμη και υπομονή. Όπως είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ΑΣΕ για ζητήματα που την αποσχολούν σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Για την Τουρκία. Όπως και όλοι οι άλλοι και η Τουρκία έχει τα ζητήματά της, ίσως περισσότερο από άλλους. ελευθερία των ΜΜΕ και η κατάσταση των δημοσιογράφων είναι κάτι το οποίο έθιξα και εγώ. Η Τουρκία είναι σημαντικός παίκτη εντό του ΑΣΕ, στο παγκόσμιο πλαίσιο. Ο Τούρκος πρέσβης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλείας του οργανισμού μας και ασχολείται με διεθνή ζητήματα και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τουρκία είναι σημαντική περιφερειακή χώρα, στην περιοχή της και γενικότερα. Οπότε ο ΑΣΕ είναι ένα καλό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει σε επαφή με την Τουρκία. πήγε σκεφτείτε τα ζητήματα του Νοτιού Καυκάσου. Η αιρεσιμότητα είναι, είναι θέμα δικό σας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΑΣΕ εγώ όταν μιλάω ως Γενικός Γραμματέας του ΑΣΕΚ προσωπώ τους 57, οπότε δεν υπάρχει για μένα αιρεσιμότητα ως προς κανέναν. Αλλά μπορεί να υπάρξει αιρεσιμότητα στη σχέση μεταξύ των χωρών, ε, οι ομάδων χωρών και οπωσδήποτε μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για να προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά βεβαίως η αιρεσιμότητα είναι και ε, δυνητικά επικίνδυνη. Και δηλαδή πρέπει να δούμε ποιο θέτει όρου σε σχέση με τι είναι στο μέσο στον οποίο θα ήμουν ε, προσεκτικός. Συμφωνώ πλήρως για τα ζητήματα πολυμερούς διπλωματίας. Ε, αν δεν τα πίστευα αυτά δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περήφανη. Μόλις έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και βεβαίω ε, θεωρώ πως ε, οι πολυμερείς σχέσεις είναι σημαντικές σήμερα για να είναι όλοι σε ένα διάλογο. Ο διάλογος όπως είπα είναι φτηνός και είναι καλό να έχουμε αυτές τις ευκαιρίες έτσι και σε καιρούς δύσκολους. Είμαστε σε καιρούς όπου οι σχέσεις μεταξύ της κοινότητας του ΑΣΕ είναι δυσκολότερες από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Οι συζητήσεις εντός του ΑΣΕ είναι πιο δύσκολες σήμερα και άρα σημαντικό είναι να ε, συζητήσουμε αυτό το, το εργαλείο διαλόγου. Τέλος, για τις εκλογές. Ε, Πράγματι έχουν τους ανθρώπους σε επιτόπου και μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα το οποίο είναι στη δική μας την ατζέντα. Δεν ξέρω καν σε ποιανού την ατζέντα είναι, αλλά βεβαίω στο πλαίσιο της εντολής μας και παραδείγματος χάρη κινούμαστε στο πλαίσιο της, ε, του ψηφίσματος υπερθμών 244. Οπότε θα πρέπει, αν είμαστε παρόντες, να έχουμε τη δική μας εντολή. Οπότε μπορεί να είναι η κατάσταση προβληματική, αλλά με βάση αυτούς τους περιορισμούς, όπως σας είπα, οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα και υπάρχει επιθυμία, αν υπάρχει επιθυμία μπορούμε να, να το εξετάσουμε, δηλαδή το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Ήταν καλή η συζήτηση. Και Βεβαίω θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για τα ζητήματα, όπως είπα, και τις παρατήρησης των εκλογών, αλλά και την συνεργασία στην οικοδόμηση θεσμικών οργάνων. Θεωρώ πως μπορούμε να έχουμε και μια κάποια άμυλα, αν θέλετε, αλλά αυτή θα έχει καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ε, ναι, ναι, ναι. Περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το 4 δηλαδή. Στρατηγική για το κέρας της Αφρικής. Πού είναι ο κύριος Τάνοκ. Πήγε μου φαίνεται σε κάποια αποστολή διερευνητική έφυγε. Ούτε η κυρία Γιαννάκου είναι εδώ. Dr. Tennant has arrived. Ήρθε ο κύριος Τάνοκ. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πριν από μια-δύο εβδομάδε έκανα μια δυο εκανα παρουσίαση για την εκθέση Εδώ τώρα θα πω κάποια σχόλια για την ε, σημερινή κατάσταση. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδου εισηγητέ για τη συνεργασία του στην επίτευξη μια πολύ ισορροπημένη έκθεση με 18 συμβιβαστικέ τροπολογίε ανάμεσα στο βασικό κορμό της ε, πολιτικής εξωτερικής, της εξωτερικής πολιτικής, ε, δηλαδή κατά πολέμηση της πειρατείας, της τρομοκρατίας, των εγκλημάτων, στην περιοχή που είναι για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της έκθεσης. Μα δεν θέλω να αγνοήσω τις υπόλοιπα, τα υπόλοιπα σχετικά θέματα ανάπτυξη ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, οικονομία και βέβαια ανάγκη για περισσότερη περιφερειακή ολοκλήρωση και το ρόλο του ειδικού ευρωπαϊκού αποστελμένου και της Αφρικανικής Ένωσης στην περιοχή. Καταφέραμε λοιπόν 18 συμβαστικές να φτιάξουμε για τα βασικά αυτά ε, θέματα. Επίσης ε, θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η μορφή της επόμενης, ε, της επόμενης κυβέρνηση της Αιθιοπίας μετά από το θάνατο του Πρωθυπουργού και το τι συμβαίνει στην Ερυθρέα αυτή τη στιγμή όπου χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όμως να σας προεκφράσω την απογοήτευσή μου κύριε Πρόεδρε για την ομάδα σας, το ΕΛΚΑ γιατί ε, ο κ. Στάντον ήταν εισηγητής ε, και ήθελε να διαγραφεί οποιαδήποτε αναφορά στη Σομαλιλάνδη και κυρίως το γεγονός ότι είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα και ακόμα και την, σημειώσουμε την επιθυμία μας να αναγνωριστεί ως κράτη. Εδώ είναι ένα πολύ βασικό θέμα εξωτερική πολιτικής για την Αφρική και δεν μπορεί να μπει στην άκρη και να αγνοήθηκε στη διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία. Η διαγραφή λοιπόν κάθε αναφορά στο θέμα αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Για όσους δεν γνωρίζουν πολλά για τη Σομαλία, να σας πω, μάλλον για τη Σομαλιλάνδη, ήταν για λίγο ανεξάρτητη το 1960 και ορισμένοι Γάλλοι συνάδελφοι ανάμεσα στην αντιπροσωπεία της, ε, στην την ε, αντιπροσωπεία στο ΕΛΚΕ προσπαθούν να προστατεύσουν ε, την Σομαλία από οποιοδήποτε ανταγωνισμό από μια ανεξάρτητη Σομαλιλάνδη. Ορισμένοι Ισπανοί ανησυχούν όσον αφορά το καταλανικό αποσχεστικό κίνημα που φτιάνει ε, αυτή τη στιγμή, αλλά η Καθαλούν είναι τμήμα της ε, Ισπανίας εδώ και 300 χρόνια. Ακόμα και αν η Σομαλιλάνδη αποσχιστεί, δεν θα αποτελέσει, νομίζω, ε, προηγούμενο σε παγκόσμια κλίματα. Ούτε θυμάμαι Ισπανού συναδέλφου από το ΕΛΚ να αντιστέκονται στην ανεξαρτησία της Ερυθρέας ή του Νοτιού Σουδάν όταν συζητήθηκαν τον περασμένη δεκαετία γιατί λοιπόν δημιουργείται τόσο μεγάλο πρόβλημα για τη Σομαλιλάνδη είναι θέμα της ίδιας της Σομαλιλάνδης να ξεκινήσει διάλογο με το Μογαντήσιο και αυτό είναι κάτι που έχει εξάλλου σημειωθεί και στηριχτεί στο τελευταίο τελικό ανακοινωθέν τη διάσκεψης του Λονδίνου οπότε καταλαβαίνετε αμφιβάλλω αν οποιαδήποτε σοβαρή έκθεση μπορεί να αναφέρει ε, που να ασχολείται μάλλον με την Ισπανία μπορεί να αναφέρει τη Σομαλιλάνδη. Ε, αυτή είναι λοιπόν η συμβιβαστική 13. Συντηρίζω φυσικά και την παράγραφο 2 της α, ε, γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. Και κατά τα άλλα θα είναι έτοιμος ο κατάλογος ψηφοφορίας για αύριο το πρωί. Έχω όλες τις υποδείξεις για τους υπαλλήλους της γραμματείας και Ελπίζω ότι έτσι θα το μπορέσουμε να το χειριστούμε. Θα μπορούσαμε ίσως για τη συμβιβαστική 13 να ψηφίσουμε το ε, συμβαστική και μετά να ψηφίσουμε χωριστά την ε, τροπολογία των Ζων για να διαγραφεί η αναφορά στη Σομαλιλάνδη και την ανεξαρτησία της. Ε, Σχόλια λοιπόν των συναδέλφων περιμένω. Αυτά έχω να πω για την ώρα και βέβαια ψηφοφορία αύριο το πρωί. Eh, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αλλά ιδίως να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ. Για μιλητής, ε, διότι ο κύριος Τάνοκ ε, εργάστηκε πάρα πολύ σοβαρά και εις βάθος, οπότε και πάλι, πάλι να ευχαριστήσω και όλους όσους έχουν συμμετάσχει πάρα πολύ καλά τα πήγαμε και και γι' αυτό αυτές οι 200 τόσες τροπολογίες χτενίστηκαν όπως πρέπει. Από πλευρά τώρα να σας πω, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα ε, να αναδείξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν είναι δυνατόν να ε, κολλήσουμε στις λεπτομέρειες, θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται ε, με τις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών χωρών, πρόκειται εδώ πέρα για κάποιο είδους ε, γενική εντολή, για κάποιο είδους ε, ε, ε δι, διάδημα, για να μπορεί κανείς να, να ζήσει με αξιοπρέπεια, με ελευθερία, όπως επιτάσσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Το αξίζει ο κόσμος αυτός το τη Αφρικής γιατί έχουν υποφέρει τόσα τόσο καιρό. Και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ γιατί λάβατε υπόψη ε, όλα όσα όλοι οι συναδελφοί επιθύμησαν. Έχουμε μας δεδομένη την εντολή για τα διαβήματα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, για τους όρους και τις προϋποθέσεις, όλα αυτά ξεκαθαρίστηκαν και ακριβώς αυτά τα οποία πρεσβεύει η Επιτροπή μας. Πάντως αυτό το οποίο είναι δύσκολο είναι να δούμε πώς θα ε, αναδείξουμε πώς έγινε εκεί η απώλεια της Θέλουμε αυτό να ληφθεί υπόψη, θέλουμε αυτό να τονιστεί, να αναδειχτεί, να προταθεί. Γιατί υπάρχουν εκεί κάποιες δυσκολίες, υπήρξαν ανέκαναν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Σαν δηλαδή εδώ πέρα, να υπάρχει ένα κενό μία φούσκα, πώς να το πούμε. Τα λέω κι εγώ στην Σουηδία. Θα πρέπει να βρούμε κάποιο είδου συμβασμό, κάποιο είδου συμφωνία. Ε, δεν μπορούσε να κατονομάσει χώρες ο κ. Τάνο βεβαίως, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, χώρες ε, περισσότερες από μία ε, έχουμε, έχουμε από διάφορες χώρες, δημοσιογράφους. Ελπίζω τελικά να διαμορφωθεί η κατάλληλη ε, πλειοψηφία, ούτω ώστε να αναδειχθούν τα θέματα τα οποία πρέπει. Έχουμε την ε, τροπολογία 34 των Σοσιαλδημοκρατών πάντως και έχουμε επίσης και τις τροπολογίες Επιτροπής Ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι σας τα είπα όπως χρειάζεται. Δεν θέλησα να ειρωνευτώ, να επικρίνω. Απλώς θα πρέπει εξ αρχής να δώσουμε το, το σωστό μήνυμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης κατά πόσον θα μπορέσουμε ίσως το κείμενο αυτό να το χτενίσουμε κάπως γιατί είναι αρκετά ογκώδες, αρκετά μακροσκελές και θα πρέπει οπωσδήποτε ξαναλέω να ε, αναδείξουν το θέμα της ε, τόσο επιθυμητής ανεξαρτησίας της χώρας. Κύριε Γκόμες, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τάνοκ διότι κατέβαλε προσπάθειες να μπορέσει να ε, κλείσει τους απρέτους ε, αναγκαίους συμβιβασμούς. Έχουμε εδώ διαφορετικές απόψεις, ε, αλλά και όπου διαφέρουμε τελικά μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και όσον αφορά το Σομάλιλαντ και τελικά συμφώνησε να μπει αυτό το οποίο εμείς του ζητήσαμε χωρίς να θεωρηθεί ότι αυτό παραβλάβει την στρατηγική του κοινοβουλίου. Επίσης, θέλουμε να μπει τελικά αυτό το οποίο έχουν ζητήσει νομίζω οι πράσινοι όσον αφορά τις εισβολές. Τις εισβολές της Αιθιοπίας στην Κένια το 11 και το 12. Αδικαιολόγητο σε αυτές οι εισβολές ε, ε, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, τα πράγματα στη Σομαλία επιδεινώθηκαν. Έτσι. Είναι απίστευτη αυτή τα κακή η κατάσταση εκεί. Mm. Mm. Όπω θα γίνει και με τη Λέιντι Άστον, μια που βέβαια γνωρίζει την κατάσταση στις χώρες. Ε, τι θα κάνει επομένω, θα, θα βρεθεί τελικά το, το θάρρος, το κουράγιο να αντιμετωπίσει τα θέματα που έχουν βγει εκεί. Γιατί εκεί έχουμε πια αυτή την σοβούσα κρίση Αιθιοπία, Σομαλία, όλων των, των γειτόνων. Εργία και την Ερυθρία βέβαια που η κατάσταση είναι τραγική από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είπα για τον κύριο αυτόν ο οποίος είναι κατά το ίμιση Σουηδάς. Ε, πάντως έχουμε πάρα πολλές, πάρα πολλές τέτοιες ε, περιπτώσεις, νεκρούς, βασανισμούς. Ε, η μεταχείριση στις φυλακές του, του, των κρατουμένων είναι, είναι απαράδεκτη τέλος πάντων. Στην Θεοπία η κατάσταση δεν είναι και πολύ καλύτερη πάντως ε, εμείς. Θεωρούμε, κάνουμε ότι είναι συμμαχοί μας, ζανάω και το καθεστώς του ε, και, και οπότε κάνουν τα στραβά μάτια. Πάντως, στο σύγχρονο 2006 η Σομαλία κατάσταση σίγουρα έχει επιδεινωθεί. Και τι γίνεται όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων Ερυθρέας Αιθιοπίας. Ούτε τι κάνουμε τίποτα μεγάλο λάθος, όπως ξέρετε εκεί πέρα ε, έχουν δεσμευτεί οι δύο χώρες να κάνουν τη σχετική οριοθέτηση προσέφηκε στο Ιδιωτικό Δικαστήριο, το οποίο απεφάσισε, η Αιθιοπία αποφάσισε να μην συμμορφωθεί με την απόφαση του Ιδιωτικού Δικαστήριου, το οποίο προσέφηκε, οπότε και αυτό μοιραία είναι πηγή πάρα πολλών προβλημάτων. Είναι δε τρομερό, είναι τερατώδε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έπρεπε να σέβεται, να τιμά το διεθνέ δίκαιο, δεν μπορεί να ασκήσει την, υπεροχή, την επιρροή του συγγνώμη, στις χώρες αυτές, αλλά κυρίως στην Αιθιοπία. Η Αιθιοπία είναι βασικός ε, αποδέκτης ε, κονδυλίων κοινοτικών. Επομένως δεν τηρούν τα υπεσχημένα, τα συμπεφωνημένα ή της Αιθιοπίας επίσης. Στη χώρα αυτή, η κατάσταση των ανθρωπίνων είναι πάρα πολύ κακή. Σας λέω μόνο ένα μόνο αυτό το όνομα. Είναι δημοσιογράφος, βραβευμένος, αναφέρθηκε στην εκθέση πολύ σωστό, αλλά όμως πρόκειται για έναν από τις χιλιάδες των νεαρών ε, ε, Ερυθρέων ε, που υφίστανται τα ίδια. Να δούμε βέβαια τι θα μπορούμε να κάνουμε με τον Ζενάου. Νομίζω υπάρχει κάποια, κάποια ελπίδα μέσω των όσων λέει και ο κύριος Τάνοκ. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία για να κάνουμε τη διαφορά στη χώρα. Να δούμε κατά πόσο βέβαια και ο νέος ε, πρωθυπουργός θα έχει την, το, το, το, το, θάρρος να προσπαθήσει να έχει μια ευρεία ε, προσέγγιση για την λύση των προβλημάτων. Γιατί λέμε τώρα για κάποια χώρα η οποία είχε άριστες σχέσεις ε, στο ιστορικό της μεταξύ δηλαδή μουσουλμάνων και χριστιανών. Και τα τελευταία χρόνια όμως η κατάσταση ε, των σχέσεων αυτών έχει επιδεινωθεί λόγω των όσων έκανε ο πρώην υποθυπός ο κύριος ε, Ζανάουι. Προσπάθησε δηλαδή να επιβάλλει τους δικούς του ηγέτες στην μουσουλμανική κοινότητα και ξέρουν ποιες είναι οι τρομερές συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο το τι ισχύει στην Αιθιοπία είναι μια κλασική περίπτωση όπου δεν εφαρμόζουμε τις αξίες οι οποίες πιστεύουμε και τα, λόγια μας τα κάνουμε έργα και κάνουμε άλλη, υπάρχει μια διαφορά τέλος, μια, μια, μια, ένα, ένα κενό, μια, μια μεταξύ πολιτικής μας ανάπτυξης και πολιτικής εξωτερικής. Προσοχή επομένως, και μιλάμε μόνο για την Αθαπία εδώ, πέρα δικηβεύεται η όλη περιοχή του Αφρικανικού κέρατος. Τάνοκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σβέντζον. Νομίζω έχετε αποσύρει μια από τι τροπολογίε και που μου ζητούσατε να χαιρετήσω την αναγνώριση του Σομαϊλάν κλπ. Ε, και τώρα κάνετε στροφή 180 μοιρών, αλλά καταλαβαίνω. Έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η πολιτική σα ομάδα. Τέλο πάντων, δεν αναφέρω το Σομαϊλάν παρά μόνο σε μία τροπολογία σε μία παράγραφο τέλο πάντων και προσπαθώ να καλύψω σοσιαλιστές αλλά και φιλελευθέρους. Και λαμβάνει υπόψη επομένω ε, τις σοβαρές αυτές ε, αποφάσεις που αφορούν το όλο κέρας Αφρικής. Τώρα, ε, όπως γνωρίζετε, είναι περίπου τα πράγματα. Το Πούντλαντ ξέρετε ότι έχει ανεξαρτοποιηθεί και θέλει να μπει στην Ομοσπονδία όταν ε, τα πράγματα προσνόταν να σταθεροποιηθούν. Κυρία Γκόμες, σας ευχαριστώ ε, που με υποστηρίζετε σε σχέση και με την ε, Συμβαστική 13 όσον αφορά τώρα την εισβολή της Κένιας στην Σομαλία. Θα μπορούσε κανείς να βρει επιχειρήματα νομικά υπέρ της εισβολής, δηλαδή προστασία των, των απαχθέντων ε, ή των υπηκών της χώρας. Κάπως έτσι έγινε. Επίσης υπάρχει εδώ και το δικαίωμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε κάποιο κράτος εγκαταρρεύσει, τέλος πάντων. Ε, διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η εισβολή είχε και κάποια δίκαια. Αλλά τόσο αυτό είναι και θέμα. Τι να σα πω, δεν είμαι νομικό που να δικαιούμαι στο διεθνές δίκαιο, αλλά ω πολιτικό. με την κυρία Άστον το, το, το, συζήτησα το θέμα των, ε, των, των συνόρων και θεωρήθηκε ότι αυτά τα οποία βάλαμε στο κείμενο συνάδουν προς τα όσα πρεσβεύει ο ΙΕ. Είναι θετικό αυτό. Επίσης είναι θετικό το να μιλούμε με μία φωνή σε σχέση με το τι θα γίνει με τα σύνορα της Ερυθρέας. Τέλος πάντων, ε, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, ε, ναι, αυτή η απόφαση που είπατε πρέπει να είναι αφετηρία μας, τέλος πάντων. Αύριο ελπίζω ότι παρά το ότι έχουμε περί τις 100 τόσες τροπολογίες που απέμειναν μετά τους συμβασμούς, δεν θα καθυστερήσει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Η κυρία Γιαννακού έρχεται. Δεν είναι. Σχεδόν εδώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα, λέγιος Μέγιος, στο σημείο υπαριθμών 5. Το σημείο 5 αφορά την ε, έκθεση ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η κυρία Γιαννάκου είναι η συγκήτρια και πρώτα απ' όλα δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία συγκήτρια. Parece que no está la señora ponente κυρία Συγγετρία δεν έχει έρθει, από ό,τι φαίνεται. Yes. Vamos a ver lo que nos indica el secretariado, si puede acompañarnos para... Μήπως ε, θέλει το λόγο πρώτα η κυρία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου λένε ότι η κυρία Γιαννακού δεν είναι ότι δεν θέλει να έρθει, απλώς έχει ένα πρόβλημα στην είσοδο, του, όπως ξέρετε έχουμε την ε, διαδήλωση εδώ έξω και οπότε δυσκολεύεται να πλησιάσει το κοινοβούλιο, οπότε γι' αυτό και υπάρχει το προβληματάκι. Τέλος πάντων, σας προτείνω να αρχίσουμε τον κύριο Βότσον, ο οποίος επίσης είναι σκιώδης συζητητής και στη συνέχεια δώσουμε το λόγο στον Ιστίν εκπρόσωπο της Επιτροπής και ας ελπίσουμε ότι στο μεταξύ η κυρία Γιαννάκου θα μπορέσει να έρθει και να δούμε μετά, θα απολύτω το λόγο προς πολιτικό νόμο, τέλος πάντων. Κύριε Βότσον, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ την καταλαβαίνω την κυρία Γιαννάκου. Ε, όλοι τώρα δυσκολευόμαστε λόγω των γεωργών και της διαδήλωσή τους να μπούμε στην, στην, στην, ε, στο Κοινοβούλιο. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γεννάκο, την απουσία τη, για την παραγωγική τη δουλειά και για την πολύ ε, ωραία συνεδρίαση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μεταξύ σκιωδών συντονιστών και με τα χαρά μου μπορώ να σα πω ότι φτάσαμε σε μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών που χαίρον μεγάλη στήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Δεν χρειάζεται να σα πω τώρα νούμερα των τροπολογιών γιατί θα δημιουργηθεί ε, ίσως σύγχυση γιατί η αρρύθμιση διαφέρει. Πάντως το βασικό είναι να τονίσουμε το εξής, ότι δηλαδή η συμβιβαστική οι συμβαστικέ μάλλον ζητούν από την, ε, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει όλους τους στόχους του, συμβου, του, κανονισμού του Συμβουλίου 389. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι νωρίτερα φέτος το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε μια αναξιολόγηση της, οικονομική της ε, οικονομικής βοήθειας που έχει χειριστεί η Κομισιόν από το 2006 και που έχει δοθεί για τη στήριξη της ενδεχόμενης επανένωσης της Κύπρου. Για αυτό το θέμα είναι αυτή η έκθεση. Το ελεγκτικό συνεδρίο συμπέρανε πως η Κομισιόν γενικά έκανε καλή δουλειά σε δύσκολες μάλλον περιστάσεις και υπό δύσκολες συνθήκες και νομίζω πως η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου αυτό το αναγνωρίζει και καταλήγει σε κάποιες συστάσεις προς την Επιτροπή για το μέλλον. Φυσικά υπάρχει αναγνώριση του θέματος της περιουσίας που επηρεάζει τις δύο κοινότητες του νησιού και υπάρχει και μια ε, έκκληση σε μια χωριστή ψηφοφορία ε, τροπολογία με συγχωρείτε, ώστε να φτιαχτεί ένας μηχανισμός με πολυετή προοπτική, ώστε να εξασφαλιστεί ο καλύτερος σχεδιασμός. Γιατί δεν ήταν, δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουμε για όλες τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Και γι' αυτό αυτές υποβλήθηκαν χωριστά. Αλλά υπάρχουν και χωριστές τροπολογίες που καλύπτουν τον κανονισμό περί άμεσου εμπορίου που είναι ίσως όχι το κυριότερο θέμα της έκθεσης, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό για την εξέβρεση μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει στο βόρειο τμήμα του νησιού να επανέλθει στην ευημερία και θα στηρίξει την ε, διαδικασία ειρήνευσης που είναι υπό εξέλιξη. Καλωσορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυρία Γιαννάκου τη συζήτηση για αυτό το θέμα με πλουραλιστικό τρόπο και προσβλέπουμε στην στήριξη όλων των συμβιβαστικών τροπολογιών με την προϋπόθεση ότι η συγγήτρια θα στηρίξει μία μικρή προφορική τροπολογία που έχουμε να προτείνουμε. Βλέπω όμως ότι έφτασε η συγχύτρια από τότε που ξεκίνησα εγώ να μιλάω και γι' αυτό καλύτερα είναι εγώ τώρα να πάψω και να την ακούσουμε εκείνη. Όντω. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Βότσον. Όντω ήρθε κύριε Γιαννάκο. Οπότε ευθύ αμέσω το λόγο για να προσθέσει την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά οφείλεται σε μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί και εμποδίζουν την είσοδο στην πλευρά αυτή. Ε, θέλω να σημειώσω από την αρχή ότι η γνωμοδότηση αυτή αφορά αποκλειστικά στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και το πώς αυτή έχει χορηγηθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ε, ότι πρέπει να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα και δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε σχολιασμούς άλλους που αφορούν στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, αφού η έκθεση αφορά στην αποτίμηση της έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου. Ε, μέσω της έκθεσης φυσικά τονίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδοτική βοήθεια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει στα πλαίσια του υπάρχοντος κανονισμού του Συμβουλίου. Από τις συζητήσεις που έκανα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ίδιο επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστούμε τον υπάρχοντα κανονισμό. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είμαι υπέρ του να, των προτάσεων που ζητούν ε, αυτό να ενταχθεί στο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Πρώτον διότι κανείς δεν γνωρίζει, θα ήταν σαν να εικασιολογούσαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και δεύτερον διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων ανά έτος. Ε, η Κομισιόν επί του θέματος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοκομπή τόνισε ότι δεν χρειάζεται multi-annual ε, perspective και ότι μπορεί να λειτουργήσει in the year by year basis. Όσο αφορά στις τροπολογίες που προσπαθούν να ανακοινήσουν το θέμα του απευθείας εμπορίου προς το οποίο το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί, το θέμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με την γνωμοδότηση και επ' αυτού του θέματος έχει τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι η νομική βάση που επικαλούνται αυτές οι τροπολογίες έχει απορριφθεί από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 18 Δεκάτου του 2010 και μάλιστα με ψήφους 18 προς 5. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανακοίνησης του θέματος. Έχουμε καταλήξει σε πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες συζητήσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές και συμφωνήσαμε ότι αυτές οι τροπολογίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Δεν ξέρω ο κύριος Γότσον ποια ακριβώς προφορική τροπολογία θέλει να κάνει. Θα το δούμε στο τέλος, αλλά ήθελα κύριε Πρόεδρε να ξεκαθαρίσω ε, ότι η υπόθεση είναι σαφής. Η έκθεση αυτή πρώτον αποτιμά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, παραμένει στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αντιστοίχου γραφείου εκεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η βοήθεια και μάλιστα έτος προς έτος. Άρα δεν είμαστε υπέρ της, του της ένταξης στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν έχει καμία σχέση με το απευθείας εμπόριο που έχει ε, απορριφθεί από το Κοινοβούλιο και βεβαίως σημειώνεται στην έκθεση, σημειώνονται ορισμένα πράγματα που αφορούν στην πρόσβαση στις περιοχές που ελέγχονται ε, από τα ε, στρατεύματα κατοχής, από ε, τις στρατιωτικές ζώνες και βεβαίως σημειώνεται και η διάθεση, η παρένεση αν θέλετε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που υπήρξαν με το διαγωνισμό για, την, για το πρόγραμμα αφαλάτωσης. Ε, αυτό είναι περίπου το σχέδιο. Δεν είναι κάτι που βγαίνει από τα όρια της, της έκθεσης του Ελληνικού συνεδρίου και φυσικά δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά στο σύνολο του προβλήματος, του κυπριακού προβλήματος ή μια έκθεση πολιτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Τώρα, πριν δώσουμε τον λόγο στον Υπουργό Επιτροπή, θα ήθελα κύριε Βότσον να μας ε, διευκρινίσετε περί ποιες προφορικής τροπολογίας πρόκειται και τι περιέχει. Βότσον, το φοβόμουν θα με ρωτήσει πρόεδρε. Όχι, δεν έχω το κείμενο εκεί μπροστά μου, δηλαδή ακριβώς τι συζητήσαμε ε, σήμερα στους φιλελεύθερους. Πάντως θα φροντίσω να το λάβει η γραμματεία μας και να το δώσει στην κυρία Γιαννάκο το συντομότερο δυνατόν. Τώρα, επίτρεψε πρόεδρε να πω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Γιαννάκο. Πρόκειτο για μία από τις συστάσεις του Νοτικού Συνεδρίου που θα έπρεπε να έχουμε σε αυτό το πολιετές πρόγραμμα ε, χρηματοδότησης για την Βόρεια Κύπρο. Καλώς κύριε Βουατσόν. Ελπίζουμε επομένω ότι συντόμω θα μας γνωστοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν το, το κείμενο και αυτή τη πολιτική τροπολογία και τώρα θα λάβει το λόγο η κυρία που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που δώσατε το λόγο στην Κομισιόν και ευχαριστούμε και την Επιτροπή Εξωτερικών που συνέταξε την γνωμοδότηση και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Γιαννάκου που συνέταξε το σχέδιο αυτό. Πρέπει να παραμείνουμε πράγματι στο θέμα αυτό και να υπενθυμίσουμε πως οι στόχοι του προγράμματος βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη με στόχο να διευκολυνθεί η επανένωση της νήσου. Σημασία έχει να τονίσουμε πως αυτή η βοήθεια είναι η μόνη βοήθεια που λαμβάνουν οι Τουρκοκύπροι που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη βοήθεια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω επίσης πως επαναλήφθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο η εμπιστοσύνη τους ε, στη δουλειά μας. Έχουν κάνει κατά την απόψή μας μια ειλικρινή αξιολόγηση της δουλειάς μας. Βεβαίως έχουν αναφέρει και αδυναμίες και η Κομισιόν έχει ήδη αρχίσει να τις αντιμετωπίζει. Έχουμε κάνει λοιπόν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τώρα την βιωσιμότητα, θεωρούμε πως το δικαστήριο το ελεγκτικό συνέδριο, με συγχωρείτε, δικαίως το έθεσε ως ένα πραγματικό και υπαρκτό ζήτημα και ε, τους λόγους που σχετίζονται με αυτό. Και υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Ένας είναι η έλλειψη διοικητικής ικανότητας από πλευράς των Τουρκοκυπρίων δικαιούχων και αυτό πρέπει να το δούμε. Και κάτι άλλο το οποίο μόλις αναφέρθηκε είναι η έλλειψη προβλεψιμότητας των κονδυλίων. Και βεβαίως, σημαντικό είναι πάντα να έχουμε κατά νου την ευρύτερη πολιτική εικόνα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά σημαντικό είναι, όπως ε, συνέστησε το ελεγκτικό συνέδριο, να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα κάπως στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο επιμένοντας βεβαίως στην ανάγκη να καταλήξουμε σε μια γενική λύση, συνολική λύση του Κυπριακού. Η Κομισιόν ήδη έχει υποβάλει συγκεκριμένες ε, προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και άρα είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε στήριξη από το Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί Μπορούμε βεβαίω να καταθέσουμε προτάσει, αλλά δεν μπορούμε από μόνοι μα να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε και την αρχή του προπολογισμού, Όσον αφορά τα ζητήματα του στόχου, του κανονισμού βοηθείας, που επίσης ε, συζητήθηκε στο σχέδιο αυτό νομοδότησης και στις τροπολογίες. Κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό να αναφερθούν όλοι οι στόχοι. Όλοι είναι σημαντικοί για να επιτύχουμε τον στόχο της δουλειάς μας, για να στηρίξουμε δηλαδή την επανένωση. Και άρα καλωσορίζουμε τις ε, τροπολογίες που αναφέρουν αυτούς τους στόχους. Να πω τώρα λίγα λόγια για το ζήτημα των ε, δικοινοτικών έργων. Όταν η Κομισιόν στην ε, απόφαση χρηματοδότησης εξετάζει το εάν και σε ποιο βαθμό θα χρηματοδοτήσει ένα έργο, μετράμε το εάν είναι έτοιμο, όριμο και βιώσιμο ένα έργο. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά δικοινοτικά έργα. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε πάντα να προτείνουμε ε, τόσα όσα θα θέλαμε. Για ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα για το έργο της αφαλάτωσης. Θεωρώ. Πρώτα απ' όλα το ελεγκτικό συνέδριο δικαίως λέει πως ε, πρόκειται για αποτυχία και πισωγύρισμα του προγράμματος. Όμως θα ήθελα να αναφέρω τις απόψεις της Κομισιόν όπως αναφέρονται στην ετήσια έκθεση της, ε, την οποία αποστέλουμε κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο, πώς το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα είχε προβλήματα, δεν τα έχουμε κρύψει, προβλήματα που αφορούσαν την πρόσβαση στο εργοτάξιο, προβλήματα πρόσβασης που επέβαλε ο τουρκικός στρατός που προέκυψαν το τέλος του 2010 και μόλις δεν υπήρχαν πλέον αυτές οι, αυτοί οι περιορισμοί ο εργολάβος δεν ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει. Επίσης αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι πως οι πιστώσεις που είχαν δεσμευτεί για αυτό το έργο Ε, έφτασαν στο τέλος του χρόνου διαθεσιμότητας, δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν εκταμιεύτηκαν, αλλά λόγω κάποιων περιορισμών ε, στα έτη χρήσης τους δεν είναι πλέον ε, διαθέσιμες. Οπότε, εάν καταλήξουμε στο ότι θέλουμε ένα τέτοιο έργο ή κάποιο παρόμοιο έργο, ελπίζουμε να μπορούμε να βασιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ε, στήριξη όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος να το πρατηθεί. Να σου πω τη δική μου άποψη, όχι ως πρόεδρος, αλλά ως εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου ε, ε, την έκθεση και η πολιτική μας ομάδα βεβαίως συμφωνεί με κάθε προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, κάτι το οποίο να οδηγεί στην επανένωση της νήσου και γι' αυτό ακριβώς και συμφωνούμε και με κάθε οικονομική βοήθεια προς την τουρκο-κυπριανή κοινότητα. Όπως ακριβώς γίνεται και με τους ε, υπηκόους της Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, Από το 1984 η μισή νήσο, τέλο πάντων σχεδόν η μισή, ε, βρίσκεται υπό κατοχή, 40.000 Τούρκου στρατιώτε και επομένω ε, έτσι δεν είναι καθόλου εύκολο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να εφαρμόσει τα όσα αποφασίστηκαν. Πρόκειται για μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και επομένω ο βασικό στόχος της ε, πολιτικής μας ομάδας είναι να μπορέσει το νησί να επανενοποιηθεί. Αυτά. Απλώ εφαρμίζω του μου και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα που να υπονομεύει κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια τη Κυπριακή ε, Κυβέρνηση για την επανένωση. Τέλο πάντων, ε, νομίζουμε ότι αυτή η βοήθεια έχει ε, καταλήξει σε έργα υποδομή, έχει βελτιώσει το επίπεδο ζωή του κόσμου, αλλά από δική μα πλευρά αυτή η οικονομική βοήθεια είναι δυνατόν να ε, γίνει επί τη βάση πολιετούς προγράμματος γιατί έτσι θα αποφύγουμε το να δίνεται ένα λανθασμένο μήνυμα ότι δηλαδή δεν ελπίζουμε να υπάρξει ε, κάποιο είδους ε, λύση στο Κυπριακό. Επομένως, έχουμε δεδομένο τον κανονισμό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους Ελληνοκυπρίους, ε, αυτούς δηλαδή που κατέχουν το, το έδαφος γη κατά 78%. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρώσουμε ε, τα όσα προβλεκονισμούς, αλλά δεν μπορούμε, διότι ο τουρκοκυπριακός, ε, ο τουρκικός στρατός μάλλον, δεν αφήνει ε, αυτού που έχουν λάβει κάποια έργα να τα εκτελέσουν. Τέλο, να πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πρώτη φράση εκεί που λέει ότι τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να επιλύσουμε το Κυπριακό, το τι θα γίνει με, με, την, ε, με τι ιδιοκτησίε, κάτι το οποίο αφορά και τι δύο κοινότητε. Αλλά έχουμε αυτή τη συμβαστική διάδεξη που λέει ότι μια επίλυξη αυτού του προβλήματο τη κυριότητα, τη ιδιοκτησία τη γη μπορεί να γίνει με κάποιο είδου γενικότερη λύση, ολοκληρωμένη λύση και όσον αφορά τα, τα, τα επόμενα, τα μελλοντικά βήματα για την ε, επανενοποίηση. Τέλο πάντων, δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε την κυρία Γιαννάκου και ελπίζουμε ε, ότι θα βοηθήσουν και οι συμβασμοί και να μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα δεν υπάρχει άλλο που ζητεί το λόγο. Α, κυρία Γιαννάκου θέλει το λόγο. Ε, για να... Κάποια συμπεράσματα να εξαγάγεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πρέπει να πω ότι επεδείχθη ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συναδέλφους και είχαμε μια καλή συζήτηση για τις ε, ε, συμβιβαστικές τροπολογίες ε, και νομίζω ότι θα καταφέρουμε και στην ψηφοφορία να έχουμε μια αποτίμηση της έκθεσης του ελληνικού συνεδρίου τέτοια που να παραμένει στο στόχο. Τώρα για το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα κύριε Πρόεδρε είναι σαφές, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για να κάνει κανείς τέτοιες προβλέψεις. Είναι κατανοητό και το έχει πει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς. Πρέπει να αρχίσει να γίνεται κάτι πραγματικά, δηλαδή να γίνει ένα έργο και να μην πάει στράφη όπως έγινε με το έργο της αφαλάτωσης και να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή είναι πάγια και δεν θα αλλάξει ή ότι δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό και γι' αυτό ακριβώς εγώ είμαι αντίθετη στην άποψη αυτή της ένταξης και από την ώρα που υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης δεν υπάρχει νομίζω κανένα πρόβλημα. Ε, κατά τα άλλα κύριε Πρόεδρε με άλλα θέματα όπως ετώνησα από την αρχή δεν πρέπει να εμπλακεί η έκθεση αυτή δηλαδή είτε με τη γενικότερη λύση του Κυπριακού είτε με τα γενικά ζητήματα είτε με κάτι που έχει απορριφθεί από το Κοινοβούλιο όπως είναι το απευθείας εμπόριο διότι τότε η έκθεση θα αποτελούσε απλώς ένα αντικείμενο συγκρούσεων και όχι μια ουσιαστική βοήθεια του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δουλειά που κάνει και με το γραφείο που έχει εγκαταστήσει ε, στην νότια πλευρά του νησιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννάκου, ο Πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο για αυτή την έκθεση και τώρα. Πάμε στο σημείο παριθμών 6, το οποίο αφορά την ενημέρωση να αφορά την ομάδα εργασίας 14 ε, Νοεμβρίου για τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα, ο οποίος εργάζεται στην ομάδα επαφής. Eh, Στο πρόεδρε, όντως έχουμε πέντε συναδέλφους με τους ε, τέσσερις τους πρώτων και που ασχοληθήκαμε ε, με τα όσα έγιναν για τη σχέση με την Αίγυπτο από την υπατή εκπρόσωπο Πρόκειται για τη συνέχιση των προσπαθειών που, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης με την Ισία και η Ορδανία και θέλουμε έτσι να στηρίξουμε τις διαδικασίες μετασχηματισμού της ε, Αραβικής Άνοιξης. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια δουλειά μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και η ε, Πατήκη Πρόσωπος συνοδεύεται επομένως από εμάς και βέβαια, ξέρετε, εμεί έχουμε τα δικά μα θέματα, τη δική μα πολιτική ατζέντα. Ε, ό,τι δηλαδή περνάει μέσα από αντιπροσωπείε, επιτροπέ κλπ. Αλλά πάντω ε, έτσι ε, δίνουμε μήνυμα ενότητα όσον αφορά τα θεσμικά όργανα τη Ένωση. Γιατί τέλο πάντων είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με την Αραβική Άνοιξη. Είπατε εκπρόσωπο, ε, ε, αναπτύσσει αυτό το έργο, είναι δύσκολο, ασχολείται και ο κ. Σταγιάννη, ο αντιπρόεδρος ο Επίτροπος ε, ε, για τα θέματα γειτνίασης, ο Γιώργος Φίλε, ε, επίσης ο Βερνατολιών, ο Ευρωπαίος Διπλωμάτης, διάφοροι επίσης υπουργοί, υφυπουργοί, έχουμε και βεβαίως την Κυπρία υπουργό που ασχολείται, το Βούλγαρος, ο Σουηδός, υπουργοί. Και επομένω με αυτόν τον τρόπο, εκτός του να εμπλέκουμε και πολιτικούς, έχουμε και πάνω από 100 Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Γιατί όπως γνωρίζετε, η Αίγυπτος δεν χρειάζεται μόνο βοήθεια στην μετάβαση στη δημοκρατία, αλλά η χώρα χρειάζεται και κάποια επάνωδο στην ανάπτυξη. Να δοθεί δυναμισμός στην οικονομία που τόσο πολύ επλήγει από τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Επομένω, είχαμε μια μερίσια διάταξη πολιτική, επιχειρηματική, οικονομική. Είχαμε διάφορους συνομιλητέ της πολιτική τάξη και της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτοί όχι μόνο εκπροσώπησαν των πολιτών και ήταν κάποιοι που τους έστειλαν οι αρχές, αλλά ήταν και εκπρόσωποι των πολιτών που ε, είχαν οριστεί ε, και από το, τη δική μας υπηρεσία, το δικό μας γραφείο στην ε, χώρα, στην Αίγυπτο. Και οι και και οι υπόλοιποι βοηθήσαμε στο να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και με συνομιλητές που δεν προχόντουσαν από επίσημα θεσμικά όργανα της χώρας. Είχαμε τους πράσινους ε, μια συνάδελφο, ε, τέλος πάντων τελευταία στιγμή αυτά καταφέραμε να κάνουμε, αλλά επίσης ε, προσχωρήσαμε αρκετά όσον αφορά ε, τον κύριο Φέλε, με του εκπροσώπιων των πολιτών. Έγινε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων επίση με την συντακτική συνέλευση, δηλαδή του Αιγυπτίου ε, που ασχολούνται με το καινούριο Σύνταγμα και επίση με την Γερουσία, ε, μια που το κοινοβούλιο έχει διαλυθεί. Επίση, με αυτή τη συντακτική συνέλευση αντιμετωπίστηκε το θέμα το οποίο τώρα έχει αναδειχθεί και συζητιέται πάρα πολύ όσον αφορά τι, την, τι θα γίνει με τα αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το κατά πόσον η Σαρία, ο Ισλαμικός νόμος θα είναι ε, η βασική πηγή δικαίου για τη χώρα. Και οι μειοψηφούντες ε, κόπτες έλεγαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία χωρίς να περάσουν από ψηφοφορία ούτως ώστε να καταλήξουν σε κάποιο σύνταγμα. Ζωντανός διάλογος, ε, και, ήταν και θέματα που μας ενδιαφέραν εκεί πέρα. Είχα μια πολύ μεγάλη μακρά συνάντηση για όλα αυτά, αλλά όπως σας είπα ήταν πολύ χρονοπτικά τα αποτελέσματα για όλες τις πλευρές. Επίσης, Πρόεδρε, θα πρέπει να σας πω ότι στον διάλογο αυτόν ε, συμμετέσχε και ο Επίτροπος Φίλε, ε, ο ειδικό εκπρόσωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριο Λαμπρινίδη, ο παλαιό ευρωβουλευτή, συνάδελφο έγινε και κάποιο δείπνο για όλους όσους ε, είχαμε δουλέψει εκεί και επίσης είχαμε συμμετοχή και των συναδέλφων σε αυτό το δείπνο εργασίας. Επίσης είχαμε την ευκαιρία στην Αίγυπτο ε, να τους εξηγήσουμε όλα μας τα, θέματα, έστω και ε, συντόμου, μα τόσοι πολλοί και έτσι είπαμε ότι τους καλούμε, καλούμε προσώπους της Αιγύπτου να έρθουν στην Ολομέλεια και μας είπαν ότι θα έρθουν. Επίσης, ε, είχαμε την πολιτική task force, ας το πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, είχαμε και task force επίσης στα θέματα τα επιχειρηματικά, τα τουριστικά, ε, ασχολήθηκε με αυτά ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη και μπορέσαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και ενδιαφέροντος και βέβαια το θέμα μας ήταν τι θα γίνει με την Ισλαμοποίηση, τι γίνεται με όλα τα θέματα που αφορούν τη θρησκευτική πλευρά της ε, Αραβικής Άνοιξης. Πατή εκπρόσωπος συζήτησε, θεωρήσαμε ότι είναι θετικά τα και αυτής της επαφής και πάντως θα πρέπει να δούμε ότι με λίγα λόγια, πρόκειτο για πάρα πολύ θετική παραγωγική συνάντηση. Ε, μια αξιοπρέπεια, με, με, με ε, δημιουργικότητα έγιναν οι επαφές μας εκεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, σχέσεις μας με την Αίγυπτο, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο όπως αυτός, αυτή η συνάντηση με, με κάποιον διαρκή και συνεπή διάλογο. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, κάνουμε το ίδιο και με άλλες χώρες της περιοχής. Πάντως ε, αυτό που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε για μια που μας έχει είναι το τι έγινε στην ΝΑΙΤΟ τις τελευταίες ε, τις τελευταίες στην Αίγυπτο τις διαδηλώσεις στην Ταχύρ και τα θύματα εκεί, την παρέτηση κάποιων ψηλών αξιωματούχων όπως του Γενικού Εισαγγελέα και πάντως όπως έγιναν και οι σχετικέ δηλώσεις μετά τη συνάντηση, είπαμε ότι εμεί προχωρούμε και τις σχέσεις μας και θέλουμε να γίνει πάρα πολύ ε, να γίνει σεβαστή από την Αίγυπτο η αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Αυτά κύριε Πρόεδρε με λίγα λόγια. τα συμπεράσματα αυτά είναι κάποια συμπεράσματα τα οποία ε, βρήκαν σύμφωνα και, τα, και τις δύο πλευρές. Βέβαια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα κατάσταση των γυναικών και των ε, μειονοτήτων που δεν ε, αναγνωρίζονται ως μειονότητες ε, από την Αίγυπτο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε ακριβώς και την παρέμβαση αυτή της, της, της βουλευτίνας από την κοινότητα των κοπτών που δεν αναγνωρίζεται. Πάντως όλα αυτά τα είπαμε, συμμετέσχουν πάνω από 600 πρόσωπα από όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Τους προσεκάλεσε όλους να συμμετάσχουν οι πρόσωπος και το σημαντικό επαναλαμβάνω είναι το ότι δώσαμε εικόνα ενότητος. Κυρία Νάης από τους Φιλελευθέρους, κυρία Ντεκάιζερ ήρθε επίσης από τους σοσιαλιστές, κύριε Σαρτζεντίνη, από τους Πρασίνους και ο κύριος Καρίμ από τους ε, συντηρητικούς ε, οι οποίοι ε, φαντάζομαι συμμερίζονται τις απόψεις που σας είπα και ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαφράγκα, έχουμε κάποιους που έχουν ζητήσει το λόγο, Κυρία Σάκη πρώτη. Σκάκι, διορθώνει. Thank you. <laughs> Sorry a little bit lost in translation, but the second time it came through clearly. Κάπως ε, δεν ακούστηκε το όνομά μου στην, στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβα. Ε, εκτιμώ την... Ε, ε, τα, τις εισηγήσει που ακούσαμε εδώ ε, για την αποστολή στην αποστολή. Θέλω, έχω πολλά μια ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο, γιατί πιστεύω πως η Task Force ε, λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αναζήτησης τερικής σχέση σε πιο ισότιμο επίπεδο και φαίνεται πως υπάρχουν πολλές ελπίδες, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και διερευνητικής φύσης εργασίες. Όλα αυτά λοιπόν στην ουσία φαίνεται να οδηγούν Ε, μάλλον να εντάσσονται στη λάβαρο του more for more, δηλαδή περισσότερα και περισσότερα ισορροπία, ε, προσήλωση στις αξίες τις οποίες ε, μας είναι μας ιδιαίτερα προσφυλής. Και ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι διαδράσεις μας στις πρόσφατες εξελίξεις του προ και τις δράσεις του Πρόεδρου Μόρση. Ήδη τίθεται σε δοκιμασία αυτή η διαδικασία more for more με την τοποθέτησή του πάνω από όλα και κάθε αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν πιστεύει ο κύριος Αλαφράγκα ε, ότι πρέπει τώρα να επαναλάβουμε τι εννοούμε με την αρχή αυτή του μορφωμόρ. Γιατί το αντίθετο, το αντίθετο είναι less for less, λιγότερα και λιγότερα. Και πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί γιατί βασικά μιλάμε στον λαό της Αιγύπτου, στην επόμενη γενεά και είναι πολύ σημαντικό να του δείξουμε πως όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται μόνο στο δρόμο, αλλά ότι στους, κατεβαίνοντας στους δρόμους ε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος μια ψήφος, είναι υποστήριξη, η λαϊκή υποστήριξη για τις αποφάσεις, αλλά και ε, θεμελίωση σε βασικές αξίες. Gracias, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρωί μιλούσα σε διπλωμάτες στο Λονδίνο για τον ρόλο του Κοινοβουλίου μας όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και βεβαίω οφείλουμε να επενέσουμε την κυρία Βαρονιάστον γιατί έφερε πέντε ευρωβουλευτές, τον κύριο Μπράιον Κρόου, ο οποίος ήταν ε, αρμόδιος ε, για τα ζητήματα αυτά, είπε πως ε, το πρότυπο στο οποίο μοιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μάλλον η Αμερικανική Γερουσία παρά η Βουλή των Κοινοτήτων όσον αφορά τον έλεγχο της υπηρεσίας εξωτερική δράση, Οπότε θέλω πάλι να ευχαριστήσω την κάθε και βεβαίως για το ότι υπάρχουν πολυμερή δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βεβαίω ε, το ζήτημά μου, το ερώτημά μου είναι πως ε, ο κύριος Μόρση έδωσε εαυτόν του ουσιαστικά ε, εξουσίες δικτάτορα, δεν μπορεί να τον αγγίξει τίποτα, δεν υπάρχει και κοινοβούλια και δεν υπάρχει και και βέβαια όταν μιλάμε για αδελφό μουσουλμάνο ανησυχώ και για τις γυναίκες και για τους χριστιανούς και για το... την ασφάλεια του Ισραήλ και θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε μια που έχετε συναντήσει τον ίδιο τον πρόεδρο πρόσφατα. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να εκφράσω τι ανησυχίε μας ε, για τα όσα έγιναν μετά από τα τέσσερα διατάγματα τα οποία εξέδωσε ο πρόεδρος Μούρση που φυσικά δημιουργούν πολύ σοβαρό ε, συνταγματικό πρόβλημα και θα ήθελα να ξέρω αν ο κύριος Αλαφράγκα στην επαφή του με τους εκπροσώπους τη συντακτική συνέλευση, αν έχουν εξετάσει αυτή την κατάσταση, αν έχουν ανταλλάξει απόψει ή αν απλώς ε, ε, έλαβαν, κατέγραψαν τα γεγονότα, αλλά χωρίς κανένα είδου άλλη ε, κίνηση. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους συναδέλφου για τι ερωτήσει του πάντω. αυτό που θέλω να πω είναι, σα ξεκαθαρίσω το εξή ότι δεν είμαι παντογνώστη και κυρίως δεν είμαι προφήτη. Σας είπα τι έγινε με την Task στην Αίγυπτο. Εκεί πήγαμε με τους προέδρους, αντιπρόεδρους, σας είπα και τέλος πάντων. Ε, ε, έχουμε και τις δεδομένες εξελίξεις που έγιναν από τότε. Πάντως, πρόεδρε, δικαιούται ο Πάσα ένας στην Επιτροπή μας να τοποθετηθεί. Πάντω αυτό το οποίο είπαμε νομίζω ότι βρίσκουμε όλου σύμφωνου στην ε, Επιτροπή μας, στην αποστολή μας και είπαμε ότι όλοι συμφωνούμε και το αναγνώρισε ο κ. ότι πήγε καλά αυτή η αποστολή και ότι το Κοινοβούλιο είναι πολύ σωστό το ότι ε, συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και, και επίσης ε, θυμάστε την προηγούμενη επαφή μας το τότε με, με τους αδελφούς και είπαμε ότι είχαμε ε, έντονη αντιπαράθεση στις, ε, στις, στην, στην συνάντηση που έγινε στη συντακτική συνέντευξη. Πάντως, υπήρξε πρόβλημα με την αξιοπιστία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είχαμε στηρίξει τον προηγούμενο ηγέτη της χώρας. Πάντως, παρουσία μας, η κινητοποίηση και όλα αυτά τα οποία οργάνωσε, οι εκδηλώσει που οργάνωσε η όλα αυτά απέδειξαν ότι θέλουμε να στηρίξουμε το μετασχηματισμό της χώρας. Η χώρα αυτή είναι πρωταγωνιστής πια, ε, όπως ξέρουμε, για την κρίση που σοβεί στη Γάζα. Κυρία Σχάκη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι βασικό στοιχείο της νέας μας πολιτικής γειτνίασης. Αυτό το more for more. Πολλά για περισσότερους. Και άρα η αρχή αυτή θα πρέπει και εν προκειμένου να ισχύσει όσον αφορά το τι θα κάνει ο νέος πρόεδρος της χώρας. Όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Θα πρέπει να υπάρξει ανεξαρτησία δικαιοσύνης, διαίρεση των εξουσιών, διάκριση γνώμη των εξουσιών. και αυτό θα πρέπει να διακρίνει επομένως, δηλαδή η αφάνεια η δημοκρατισμός, όλες τις εκφάνσεις, όλες, όλους τους τομείς της διακυβέρνησης της χώρας. Είπαμε, χρειάζεται συνένεση, θα πρέπει να συνταχθεί, να εγκριθεί το Σύνταγμα, να περάσει και από δημοψήφισμα, οπότε και μετά μπορούν να γίνουν εκλογές στη χώρα. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μία μεταβατική διάταξη του συντάγματος που ορίζει ότι είναι τετραετής η εντολή και η θητεία του Πρόεδρου Μόρση. Άρα, μετά την κύρωση του συντάγματος και τις εκλογές, δεν θα γίνουν εκλογές για νέο πρόεδρο. Και θα μείνει στη θέση του ο πρόεδρος μέχρι να εξαντλήσει τη θετία, την τετραετία. Η κοινωνία των πολιτών και διάφοροι από τους με τους οποίους μιλήσαμε, για απαντήσω ο κύριο Τάνοκ και για σας εσάς κύριε πρόεδρε, είπαν λοιπόν ότι κέρδισαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι για διάφορους λόγους. Πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η δαιμονοποίηση του προηγούμενου καθεστώς. Ε, τους υποστηρίζουν διάφοροι μη προνομικοί της χώρας και είναι και οργανωμένοι σαν παράταξη αφορέας. Πάντως, όλος ο κόσμος παρακολουθεί την εξέλιξη στη χώρα, την εξέλιξη του μετασχηματισμού, δύσκολη επίπονη διαδικασία και επίσης ε, ελπίζουμε να να δρομολογηθεί η θεσμική εξέλιξη που θα βοηθήσει στην κατοχή των δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή πάντως ε, έχουμε προβλήματα, ε, εξού και οι σχετικές διαδηλώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να προσεχθούν. Σας παραπέμπω επομένως στα συμπεράσματα της Tax Force, όλα αυτά ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης άμεσων επαφών μεταξύ Αιγυπτίων και της κυρίας Άστον η οποία έλαβε υπόψη τις ευαισθησίες των κρατών μελών που εκπροσωπούνται εκεί από τους υπουργούς τους. Ήταν ξεκάθαρο το τι θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Επομένως, Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα συμπεράσματα αντικατοπτρίζουν τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Δεν επέβαλαν τα κράτη-μέλη αυτό που ήθελα στις σχέσεις μας με την ε, Αίγυπτο. Πάντως, εκτός από τα άλλα, καλύφθηκαν και οι... τα όσα ήθελαν οι τα κρατη που εκεί. Τώρα, όσον τα δικαιώματα, το είπαμε και, και αναφέραμε ιδίω το δικαιώματα των γυναικών στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Είπαμε επίση ένα άλλο θέμα ήταν το κατά πόσο θα είναι βασική πηγή δικαίου ε, η Σαρία και επίση τα δικαιώματα των, ε, των, ε, των μειοψηφιών. Τέλος πάντων, εμείς θα, θέλουμε να λάβουμε υπόψη τις, το τι ε, ε, τι έγινε με, την, με, με τις όλες εξουσίες που έχει τώρα συγκεντρώσει ο πρόεδρος και γιατί χρειάζεται, επομένως είπαμε, μια μεταβατική περίοδος όντως για να φτάσουμε στον εκδημοκρατισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκτροπή, εκτροπή όσον αφορά τη συγκεντρώση των εξουσιών και αυτό σίγουρα είναι ένα καμπανάκι κινδύνου το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα για τι τόσο ολοκληρωμένε πληροφορίε και ενημέρωση που μα κάνατε. Τώρα θα έρθει να προεδρεύσει και πάλι ο κύριο Μπροκ. Πάντω εγώ για να έχουμε αυτό το την μετάβαση των εξουσιών να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, την κατάσταση στην Γάζα. Νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί είχαμε βεβαίως, το είχαμε γράψει στην ημερήσια διάταξη πριν από την κατάπαυση του πυρός, αλλά τώρα μπορούμε να συζητήσουμε και τις πολιτικές επιπτώσεις και θα έλεγα πως ε, σε κάθε συνεδρίαση θα έπρεπε να έχουμε λίγο χρόνο να συζητάμε τα επίκαιρα θέματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τις ομάδες λοιπόν να κάνω προτάσεις για το ποια θέματα θέλουν να συζητάμε. Γιατί ασχολούμαστε με εκθέσεις ε, που έχουν προγραμματίσει εδώ και μήνες ε, και δεν έχουν μεγάλη σχέση με την επικαιρότητα. θεωρώ πως να έχουμε μία ώρα να συζητάμε την επικαιρότητα. Όχι για κάποιο ψήφισμα, απλά για μία συζήτηση για τα θέματα. Νομίζω πως θα ήταν σωστό κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Βλέπουμε λοιπόν πως η κατάσταση στη Γάζα έχει πολλά επίπεδα. Είχαμε βεβαίως την ε, άμεση αφορμή. Μετά είχαμε τις ε, ρουκέτες του Ισραήλ. Κάθε χώρα διεκδίκησε το δικαίωμά της ε, στην αυτοάμυνα. Ε, βεβαίως γνωρίζουμε και το περιβάλλον στη Μέση Ανατολή και γνωρίζουμε πως σταμάτησε αυτή η σύγκρουση, αλλά το γενικό πρόβλημα η αιτία δεν έχει εκλείψει. και ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει και η ειρηνευτική διαδικασία. Και εγώ θεωρώ πως αυτό είναι και προς το συμφέρον του ιδίου του Ισραήλ. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει με το αντιπυραυλικό σύστημα το Iron ε, τα πάντα. Βεβαίως, Ευτυχώς ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο κύριος Μόρση, μαζί με την Αμερικανική Υπουργό Εξωτερικών κατάφεραν μια κατάπαυση του πυρός. Και ταυτόχρονα βλέπουμε πως ε, αμέσως μετά από αυτό υπήρξε μια ε, απόφαση που δίνει απόλυτες εξουσίες ε, στον Αίγυπτο πρόεδρο. Βλέπουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον ε, της περιοχής. Εάν δούμε την πιθανή αστάθεια από τους ε, πρόσφυγες γιατί πάνε πρόσφυγες από την Τουρκία από την Συρία στην Τουρκία αλλά έχουν πάει διπλάσει στην Ιορδανία και βλέπουμε οικονομικά και ανθρωπιστικά προβλήματα και οδηγούμαστε σε μία αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Γιατί, εντάξει, παρόλη την κριτική που μπορεί να ασκήσει κανείς στην τα κτλ. Είναι πάντα χώρες οι οποίες έπαιζαν έναν ρόλο πιο μετριοπαθή και έχουμε τώρα τις εξελίξεις που γνωρίζετε στην Συρία και έχουμε άλλο ένα παράγοντα ανασφάλειας και βλέπουμε πως πιθανώς ακόμα και παρά τα εσωτερικά της Αιγύπτου και της Ιορδανίας γίνεται όλο και πιο δύσκολο η διεθνής κοινότητα να είναι σε θέση να εμποδίσει ε, το λαθρεμπόριο όπλων προς την ε, Γάζα. Το είχαν προσπαθήσει και πριν από τρία-τέσσερα χρόνια με την τελευταία αντιπαράθεση και το αποτέλεσμα δεν ήταν και πολύ καλό. Και άρα γίνεται δυσκολότερο μετά να πούμε και στο Ισραήλ ε, να αυτό συγκρατηθεί. Γιατί δεν κάνει τίποτα η διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τα όπλα που πάνε στη Χαμάς στη Γάζα δηλαδή, ούτε στη Χισμπολά στο Λίβανο. Και άρα αυτοί οι οποίοι είναι σκληροί αν θέλετε επιβάλλουν τη θέλησή τους και βεβαίω δεν μπορεί έτσι να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Και βέβαια αυτό θα αποτελέσει και σημαντικό θέμα στις Ισραηλινές εκλογές. και δεν υπάρχει λοιπόν και ετοιμότητα για μια ειρηνική λύση. Ταυτόχρονα βεβαίως το Ισραήλ προχωράει σε επικισμούς ε, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και αυτό οδηγεί σε ανασφάλεια προς την άλλη πλευρά και εδώ πέρα υπάρχει και το όλο ζήτημα του Ιράν και το τι θα γίνει στη Συρία και οι σχέσεις με τη Χαμάς και τη Χεσμπόλα. Ε, έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο πλέγμα που ξεκινάει από το Ιράν και φτάνει μέχρι τον ιδιαίτερο ρόλο του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας που δεν ξέρουμε αν οδηγούν στη δημοκρατία ή στη χρηματοδότηση της μη δημοκρατίας και των φονταμεταλιστών. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση συνολική η οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολη και ανησυχητική και βλέπουμε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιδράσει. Αν δούμε βεβαίως και το αίτημα του πρόεδρου Αμπάς να γίνει να αλλάξει το καθεστώς ε, μη κράτους μέλους στον ΟΗΕ και δεν ξέρουμε θα γίνει στο πλαίσιο του κουαρτέτου ή και εκτός του κουαρτέτου και αν μπορούμε να είμαστε μια αξιόπιστη ειρηνευτική δύναμη. Είναι λοιπόν δύσκολη η κατάσταση και από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι τώρα που ολοκληρώθηκαν οι Αμερικάνικες εκλογές απουσίαζε η Αμερική αλλά και πάλι εδώ πέρα στην κατάπαυση του πυρός δεν υπήρχαν Ευρωπαίοι. Όλα αυτά έγιναν χωρίς εμάς. Οπότε θεωρώ πως είναι συνολικά προβληματική η εξέλιξη. Και δεν νομίζω από καμία πλευρά να υπάρχει μια ικανοποιητική προσέγγιση. Και εγώ βεβαίως παραδοσιακά ήμουν πιο κοντά στο Ισραήλ και θα ήθελα να πω πως μπορούν να προκύψουν ουσιαστικές ψυχολογικές αλλαγές. Η Χαμάς και η θα μπορούσαν, αν το ήθελαν, να φτάσουν ε, με τις ρουκέτες ε, την Ιερουσαλήμ και το Τελαβίβη. Αν ήταν πιο ακριβείς στην στόχευσή τους, θα υπήρχαν βεβαίως και περισσότερα προβλήματα. Εάν δεν μπορούν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους ε, μόνο τους στο σχολείο, αυτό αλλάζει την ψυχολογία Ενό ολόκληρου λαού. Δηλαδή αυτή η προσωπική ανασφάλεια που μπαίνει μέσα στην οικογένεια σημαίνει είτε αποσταθεροποίηση είτε ακόμη περισσότερο σκέφτονται το, το τείχος και το πώς θα θωρακιστούν. Και τα δύο αυτά θα ήταν άσχημα. Ελπίζω να κάνω λάθος και θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας την άποψη. Για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. μπορείς μια έκθεση, ένα ψήφισμα θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Βάτσον. Oh, chairman, no. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μη εκλεγμένο σώμα είναι η Βουλή των Λόρδων, όπου και μάλιστα εκεί δεν θα ήθελα να βρίσκομαι. Δεν είμαι Λόρδος. Ε, πρόεδρε, αυτά που είπατε αντικατοπτρίζουν αυτό που πολλοί από μας πιστεύουμε σε σχέση με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί αυτή τη στιγμή 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 10 μέρες από την πλευρά των Παλαιστινίων. Ο μόνος ε, αρχηγός ήταν ο Αχμάντ Τζαφάρη και, σκοτώθηκε την πρώτη μέρα μάλιστα. Οπότε αναρωτιέται κανείς ποια είναι η αιτιολόγηση για τις συνεχιζόμενες μαζικούς βαρδαδισμού. Η Γάζα πριν από λίγο καιρό σε μια επίσημη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε ως μια ζωντανή κόλαση. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρόφιμα ή βασικά είδη επιβίωσης, δεν υπάρχει ελευθερία μετακίνησης, χρειάζεται άδεια σχεδόν για τα πάντα από τις Ισραηλινές αρχές. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες όχι μόνο έχουν γίνει ε, επιθέσεις κατά ε, πολιτών, όπλων πολιτών, αλλά πολύ συχνά πρόκειται για βομβαρδισμούς και μάλιστα βραδινούς, νυχτερινούς που θέτουν το 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυτή την ε, πολύ ε, πολυπληθή περιοχή να τρέμουν για τη ζωή τους. Δεν βλέπω κάτι που να μπορεί να αιτιολογήσει αυτή την παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σίγουρα δεν έχει καταστρέψει την αμάζη. Ίσως μάλιστα το αντίθετο αποτέλεσμα να είχε, να την κατέστησε πιο ισχυρή μακροπρόθεσμα. Αλλά πιστεύω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να γνώμε το γεγονός ότι αποτύχαμε και ότι οι Αμερικανοί απέτυχαν να προοδεύσουν για μια λύση δύο κρατών που θα μπορούσε να φέρει μια διαρκή ειρήνη. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ελάχιστα κάνει αυτή τη στιγμή. Και δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και με τις καλύτερες προσπάθειες της ΕΠΑ, της εκπροσώπους, ότι και εμείς κάνουμε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Και εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την αρκετά ανώμαλη κατάσταση όπου οι ε, Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αμερικανικά όπλα για να καταστρέψουν παλαιστινιακές υποδομές τις οποίες έχουν πληρώσει οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Αποδήποτε αλλού αυτό θα θεωρείται ως πόλεμος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Αυτό που με ανησυχεί δε περισσότερο, Πρόεδρε, είναι ότι αυτό είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ. Πολύ επικίνδυνο για το Ισραήλ γιατί υπάρχει αυξανόμενη ε, οργή και απόγνωση στο λαό της Λωρίδας της Γάζας αλλά και ε, εξοργίζονται και Άραβες γενικότερα. Ε, υπάρχει γενική καταδίκη για το τι κάνουν οι Ισραηλινοί και αλλού στον κόσμο και άρα όλο και λιγότερη υποστήριξη για τους Ισραηλινούς πράγμα το οποίο θα τους δημιουργεί προβλήματα με την αραβική μειονότητα που ζει στο κράτος του Ισραήλ το ίδιο. Ο αμυντικό δε του Ισραήλ είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ότι ο προπολογισμό των τεσσάρων Αράβων γειτόνων του. Αλλά το Ισραήλ θεωρεί, όπως θεωρούσε και ο Ναπολέοντας, ότι όσο και να ξοδεύεις δεν αρκούν από τη στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ειρήνευση πνεύμα είναι πολύ πιο ισχυρό από το σπαθί, από το ξύφο. Η κατάσταση όμω δεν είναι μόνο επικίνδυνη για το Ισραήλ, είναι και επικίνδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα είναι και περισσότερο από την αρχή τη Αραβική Άνοιξη, προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε τι σχέσει μα με άλλε χώρε στην περιοχή. Και ωστόσο το βασικό πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις της ε, προφανώς μας στήριξης για το Ισραήλ και έλλειψης ε, προφανούς στήριξη για μια γρήγορη λύση θα καταστήσει όλο και δυσκολότερο για μας ε, την θέσπιση σχέσεων με αυτές τις χώρες που, θα χρειαστούμε και θέλουμε. Και γι' αυτό πιστεύω, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να παροτρύνουμε την, επό... την είπατε εκπρόσωπό μας ε, να συζητήσει άμεσα με, όποιος και αν είναι, με όποιον και αν είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, τουλάχιστον να αναγνωρίσουν ότι αν η Αμερική δεν σκοπεύει να προβεί σε δράση, αν κατά κάποιο τρόπο αποσύρεται και αφήνει το πρόβλημα στη μοίρα του, ότι δεν θα αντισταθούν σε μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο θα έχει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη και να πάψουν πια αυτές οι φρικτές εχθροπραξίες που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρος. Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ εύστοχη η εισήγηση όσον αφορά τα προβλήματα στη Γάζα. Ακριβώ ε, όπω ε, έχουν ε, αποτυπωθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Όπω πολύ ωραία τα είπε ο κύριο Βότσον, επομένω, είναι σαφέ ότι Πρόεδρε, πρόεδρε, κοιτάξτε. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παραστώ σε αυτά που συζητήσαμε προηγουμένω όσον αφορά. Ε, που δεν μπόρεσα να είσαστε εδώ, μάλλον εσεί κύριε Πρόεδρε, όταν είπαμε για την Αίγυπτο που είχαμε τόσο, τόσο, τόσο θετικά αποκοιήματα. Όμω συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, ότι εν προκειμένου και όσον αφορά την κρίση τη Γάζα, δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να δραματίσει εκείνο τον ρόλο που τη αναλογεί. Παρ' όλα αυτά όμω μπορέσαμε να έχουμε κάποιο είδου παρέμβαση, ίσως όχι την αρίστη, αλλά τόσο είχαμε ε, καλή επικοινωνία με τον κύριο Μόσιν και στην ΕΙΤΟ ΕΕ, πέραν από τα από τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε τρεις ε, προσώπους του, ε, του, του, του Προέδρου είχαν σε σαν πρωτόκολλο βρισκόταν σε τάξη πρωθυπουργού και αλλά ήταν υψηλού επίπεδου η εκπροσώπηση τέλος πάντων ε, είχαμε την Χίλαρη Κλίντον η οποία ταξίδεψε, πήγε εκεί και ε, μπόρεσε να είναι στην καρδιά των προβλημάτων και μίλησε με τους διάφορους εμπλεκομένους οπότε ανέκτησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο η Αίγυπτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για κάθε 10 ευρώ τα οποία εξοδεύει για την ειρήνη, ταξίδευε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμως ακόμα δεν έχουμε μπορέσει να έχουμε επίδραση στα πράγματα όσο θα έπρεπε και τέλος πάντων να έχουμε το ρόλο που μας αρμόζει. Το κουαρτετό πάντως ε, έπαιξε το ρόλο που ελπίσαμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Αραβική Άνοιξη επισκέσε το Μεσανατολικό και όντως, κύριε Βότσον, η ομιλία του πρόεδρου Ομπάμα μόλις από τα καθήματα στο κάρο αυτό ε, σημαίνει ότι θα ασχοληθούν περισσότερο οι ΗΠΑ με το πρόβλημα. Τέλος πάντων, όμως τι θα γίνει με το Ιράν και τα πυρηνικά οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν την Χαμάς και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές είπαμε ότι έχουμε τις εκλογές, ε, το κόμμα του κ. Νοτανιάχου και επίση έχουμε τις διάφορες άλλες ε, πρωτοβουλίες της Βουρκής Ένωσης. Είχαμε εκεί ε, την επίσκεψη γερμανική, την γαλλική. Οπότε όλα αυτά, οι επαφέ με τον κ. Νετανιάχου σημαίνει ότι θα ξανασχοληθούμε με το πρόβλημα Επίσης, σε σχέση και με τον, τον κύριο Γκαμπρίτσι, έχω να σας πω κάτι που είπατε και εσείς πρώτα, δηλαδή να δούμε πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους μετριοπαθείς. Διότι την ε, σεμάνα αυτή πρόκειται να εκδοθεί κάποια απόφαση της Γενικής Συνέλευση όσον αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Ε, όσον αφορά το, το, το, το στον, στον ΑΕΑ. Και επίσης, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έχουμε πει ότι θα είναι κακό για την αξιοπιστία μας μετά από τόσο επιτυχείς κινήσεις όπως είπαμε για το Κάιρο, μετά από μόνο σε αυτές τις επιτυχίες να μην μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση ούτως ώστε να μπορέσουμε να, να, να αναδείξουμε το ρόλο μας, να είμαστε δυνατοί συνομιλητές για, για αυτό το πρόβλημα στο οποίο μας, μας, μας βλέπουν κάτι σαν ερυθρό, ερυθρό σταυρό που απλώς υπογράφει τα, τα τσέκ της επιταγής για τα κονδύλια. Αυτό αφορά και τη Γάζα φυσικά. Τέλο πάντων, πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα. Θα πρέπει επ' αυτού να μπορέσουμε να δούμε πώ θα κινητοποιηθούμε, τι θα γίνει εκεί μέσω τη ε, της, της ε, εκπροσώπου και γι' αυτό και εμείς επομένως να σταματήσουμε απλώς να, να, να είμαστε αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά αλλά θα πρέπει να ε, συμμετάσχουμε εκεί και σε πολιτικό επίπεδο πέραν του, του, του, του πολιτικού του βιομηχανικού κλπ. Επομένω, έχουμε το, κείμενό μα το οποίο αυτό είναι μια απαρίθμηση καλών προθέσεων. Αλλά ξαναλέω ότι είναι, είναι κατατμημένε οι προσπαθίε μα. Θα πρέπει να, να κινηθούμε κάπω αλλιώ. Και οπότε ε, να δούμε ποιε είναι οι πρωτοβουλίε τη εξωτερική ε, υπηρεσία, ε, τι κάνει η κυρία Άστον, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο όπω θέλουμε, όπω φιλοδοξούμε. Και επίση να εναρμονιστεί, ε, να, να βρεθεί μια κοινή θέση και όπως είπαμε να υποστηρίξουμε τους ε, μετριοπαθείς. Ευχαριστώ. Ο Γκαμπρίτσι είναι εδώ και άρα θα είναι σωστό να του δώσουμε το λόγο και έτσι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι όταν θα λάβουν το λόγο να, έχουν, ε, να ξέρουν, να έχουν υπόψη στη θέση του κύριου Γκαμπρίτσι. Έχετε το λόγο κύριε. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Σαλαφράγκα. Κάθε φορά που συναντιόμαστε μου θέτει τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που γίνεται. Θα ήθελα σύντομα να κάνω κάποιες τρεις παρατηρήσεις από την πλευρά της εξωτερικής υπηρεσίας. Η πρώτη είναι βέβαια ότι μπορεί να εκφράζουμε τη λύπη μας για το ότι στα όσα έγιναν η Ευρώπη δεν ήταν πιο ορατή λοιπά Αλλά πιστεύω πως η κυρία Άστον δεν εφίστη προσπαθειών κατά τη διάρκεια των, της υπόθεσης αυτής σε όλες τις επαφές που είχε με όλα τα τμήματα, τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους, τους υπόλοιπους, τον Αραβικό Σύνδεσμο κτλ. Αλλά υπάρχουν όρια πρέπει να πούμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εξωτερική εξωτερική πολιτική που εξαρτώνται γενικά από την ε, κατάσταση. Δεν εξαρτώνται από την ε, καλή θέληση, τη βούληση δράση τη εξωτερική υπηρεσία, αλλά πάντω ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει έγινε σε αυτή τη φάση που οδήγησε στην ανακοχή. Δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω και ανεξάρτητα δεν θέλω να προσθέσω κάτι στην ανάλυση του Προέδρου και του κυρίου Βότσον που είναι ιδιαίτερα διαυγής και ξεκάθαρη. Το αναγνωρίζουμε τα στοιχεία και τα βασικά, αλλά θα ήθελα να πω κάτι, μια, μάλλον κάνω μια παρατήρηση για την ανάγκη να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, αυτή τη νέα κατάσταση, γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία. Αυτή η ανακοχή, εάν τεθεί εφαρμογή θα πρέπει να οδηγήσει στο νέο άνοιγμα της γάζες, Γιατί έχουμε επιμείνει ότι το μπλοκάρισμα της γάζες το είναι, ήταν απαράδεκτο, το έχουμε καταδικάσει πολλές φορές και τώρα πιστεύω πως θα πρέπει σύντομα να σκεφτούμε και ήδη το κάνουμε για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε πρακτικά από την ευρωπαϊκή πλευρά για να ε, είμαστε χρήσιμοι και να συμβάλλουμε στην πρακτική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και το άνοιγμα και την ανάκαμψη την κοινωνικο-οικονομική της Γάζας ε, εξασφαλίζοντας βέβαια και τις ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια κτλ. Είναι μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω γιατί είναι σαφές και είδαμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά τώρα θα πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε πιο θετικοί και να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που μας δίνουν αυτή η νέα κατάσταση. Τρίτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω και σχετίζεται περισσότερο με τα όσα είπε ο κ. Σαλαφράγκα και ίσως εδώ είναι πιο εύκολο να απαντήσω γιατί δεν ψηφίζουμε η εξωτερική υπηρεσία τα κράτη-μέλη ψηφίζουν, οπότε εξαρτώμεθα από εκείνους. Πάντως, υπάρχει εδώ και κάποιο χρόνο, έχουμε συμμετάσχει στο Συμβούλιο για όπου η κυρία Άστον έθεσε επιτάπητο σε αυτό το θέμα και βεβαίως δεν απέτησε από όλου να πούν την γνώμη τους αν ήταν υπέρ κατά, αλλά επέμεινε στην ανάγκη ε, διασύνδεσης ανάμεσα σε εμά και τα μέρη, ώστε να δούμε πώς θα υπάρξει μια νέα γραμμή, μια κοινή γραμμή, γιατί είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητά μας και η ευρωπαϊκή μας η αξία θα είναι λιγότερη αν είμαστε διχασμένοι. Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζω ότι υπάρχουν επαφές ε, που είναι υπό εξέλιξη, γίνεται συζήτηση για το πώς θα ε, συνεχίσουμε και στο ΠΕΣΕ αύριο. Αυτό μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για μία μόνιμη ανησυχία. Να θέλουμε δηλαδή να βρούμε αυτή την κοινή θέση, αλλά θα είναι ε, όντως δύσκολο. Ε, θα το δούμε και εξαρτάται, όπως σας είπα, από τα κράτη-μέλη. Η ε, κυρία Νέιτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να σας... Ε, κυρία Γκόμες, με συγχωρείτε. Ε, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο εκθέσατε τα πράγματα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απόψεις της ομάδας μου και στο ψήφισμα που υιοθετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ικανοποιηθήκαμε ιδιαίτερα για το ότι για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο παίρνει μια θέση υπέρ ε, της ε, ύπαρξης Παλαιστινιακού κράτους και ελπίζω να μας ακολουθήσει και το Συμβούλιο σε αυτή τη γραμμή που ε, ακολουθήσαμε, χαράξαμε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση αυτή όχι μόνο για την κλιμάκωση αλλά για την καταπίεση την γενικότερη του Παλαιστινιακού λαού. Η Γάζα είναι μια υπαίθρια φυλακή. Αλλά προφανώς ε, η καταπίεση αυτή γίνεται αισθητή και στη δυτική όχθη και βεβαίως οι επικισμοί είναι μια πολύ επιθετική στάση του Ισραήλ. So... Δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε περισσότερο εξευτελισμό. Ε, τα γνωστά, καταθλιπτικά και επικίνδυνα. Βέβαια, ανησυχούμε και για την ασφάλεια του Ισραήλ. Και δεν θεωρούμε πως ε, έτσι όπως δρά το Ισραήλ έχει βελτιωθεί η ασφαλειά του. Αντιθέτως, ειδικά γιατί το περιβάλλον έχει επιδεινωθεί με τη σύγκρουση στην Συρία και βεβαίως το θέμα αυτό δεν αφορά την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, αλλά μπορεί να αποτελέσει το θέμα αυτό σε οποιαδήποτε αραβική χώρα. Και θεωρώ πράγματι ότι το να τηθεί προτεραιότητα η αναγνώριση που ζητάει από τον ΟΗΕ η Παλαιστίνη είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρουμε βεβαίω πως δεν ψηφίζει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι ΛΕΔΙΑΣΤΟΝ ε, μπορούν να ε, κινητοποιήσουν τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω λοιπόν η άστο να μην φυστεί προσπαθειών για να βοηθήσει το κάθε κράτος μέλος. Γιατί αυτό έχει κρίσιμη σημασία για να αποκτήσουμε ξανά μια ορμή στην ειρηνευτική διαδικασία γιατί για διάφορους λόγους ξέρετε πως είπα είναι κάπως απόμακρες αλλά και χάρη στις ΙΠΑ βεβαίως ε, ε, είχαμε την κατάπαυση του πυρός. Γιατί είδαμε αμέσω πως κινητοποιήθηκε ο πρόεδρος Ομπάμα, επικοινώνησε με τον πρόεδρο Μόσερη, έστειλε την ε, Υπουργό Εξωτερικών του και δικαίως βεβαίως θεωρείται πως αυτός σταμάτησε την επιδείνωση της κατάστασης. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό που πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. για τις ε, πιθανές αλλαγές ε, που θα μπορούσε να επιφέρει ο πρόεδρος Ομπάμα είναι μια ε, Μέση Ανατολή ελεύθερη από πριν. Αυτό σχετίζεται και με το Ιράν αλλά και με τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Εγώ ανησύχησα για το ότι πέταξε μία επανδρομένο αεροσκάφος πάνω από την Τιμόνα πρόσφατα. Δεν νομίζω πως μπορούμε να... Κανείς να μπορεί να mm. αντιληφθεί τη σημασία αυτού του γεγονότος ε, στο mm. σωστό βαθμό. Για όλους του και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. να επιτύχουμε μια Μέση Ανατολή χωρίς ε, πυρηνικά. Αλλιώς η εναλλακτική λίστα είναι ανεξέλεγκτη. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε με το Ιράν τέλος να πω πως άκουσα αυτά τα οποία είπε ο Γκραν Βάτσον και θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα και δεν χρειάζεται να ζητάμε τίποτα από τις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ έχουν τη δική τους λογική, τη δική τους σχέση με τα μέρη. εξαρτήτως του τι θα γίνει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα στη γειτονιά και μας ενδιαφέρει άμεσα το τι θα γίνει, να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. και να επιληφθεί το ζήτημα με τρόπο ουσιαστικό, όχι όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Πολλά είπαμε και στο Στασβούργο, αλλά και σήμερα. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε τις ΗΠΑ αλλά και την ε, Αίγυπτο για την ε, ανακοχή, την κατάβαση του πυρός. Αλλά το θέμα είναι τι κάναμε εμείς. Όντως, ε, μάλλον θλιβερά, θλιβερή θα είναι η απάντηση. Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Νετανιάχου γιατί πρόκειται για μια ε, απόφαση με πολιτικό κόστος το να δεχθούν επομένως και το κόμμα του να μπορεί να δεχθεί αυτή την κατάβαση του πυρός. Πολύ. Θεώρησαν ότι, να, η ευκαιρία να εισβάλλουν στη Γάζα και να, έτσι να σταματήσει η Χαμάς να εκτοξεύει τους πυράβλους. Σοβίδες τους και οπότε είχαμε πει ότι πρόκειτο ευχή να γίνει καταφύγιο τρομοκρατών αλλά κλείσανε τώρα αυτές οι ε, κλείσαν πολλοί από τους οπικισμούς εκεί αυτή η αναγωγή, η, ανα, ανακοχή ελπίζουμε ότι θα κρατήσει. Βέβαια, με την ανακοχή θα αναδιοργανωθεί, θα αγοράσει όπλα η Χαμάς. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον ε, Σερ Γκρέαμ και με την Άννα Γκόμες, όπως και όλοι συμφωνούμε, ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να κάνει κάτι ο Ομπάμα σε αυτή τη δεύτερη θητεία του. Να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες που να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια λύση που θα εμπλέκει δύο ή τρεις. Να σταματήσει να υπάρχει η δικτατορία της Χαμάς. Όντως στη Γάζα είναι κατάσταση απελπιστική, αλλά δεν είναι μόνο θέμα Ισραηλινής καταστολής. Μίλησαμε και με τον Κύπριο Υπουργό. Είχαμε όλους αυτούς τους ε, συνοπτικές εκτελέσεις της Χαμάς πριν από ένα δεκαήμενο. Και δεν θυμάμαι κανείς αυτό να το κατεδίκασε. Κανείς δεν προκάλεσε κάποιο κατεπήγον ψήφισμα. Επομένως, πολλοί κάνουν στραβά μάτια για τα εγκλήματα που γίνονται στη Γάζα από τους Άραβες κατά των Αράβων. Κύριε Μπροκ, είναι σημαντικό το πρόβλημα. Τώρα Ουσιαστικά αυτό είναι πόλεμο φθορά. Δεν ξέρω τώρα πού θα πάει αυτό. Όποιος βρει εκεί κάποια λύση, αξίζει ένα Νόμπελ ειρήνης πολύ πιο σημαντικό. Το αξίζει πολύ περισσότερο από τον Νόμπελ που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σας ευχαριστώ. Θα παει αυτο Όποιο βρει εκει καποια λυση αξιζει ενα νομπελ ειρηνη πολυ πιο σημαντικο το αξιζει πολυ περισσοτερο απο το νομπελ που πηρε η ευρωπαικη ενωση σας ευχαριστω θα ηθελα να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση χωρίς να επαναλάβω ε, τα όσα υπόθηκαν ήδη. Ωστόσο, θα αναφέρω και κάποιες εκφράσεις ε, ε, που χρησιμοποίησαν οι προλαλήσαντες γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Κάποιος είπε ότι η Γάζα είναι μια φυλακή. Αν όμως όντως είναι έτσι, τότε θα πρέπει να τα πούμε ε, ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι, φυλακοί, φύλακες είναι οι αμάς που κρατά άοπλους. Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία γιατί υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί με τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί ε, κινδυνεύουν από βομβαρδισμό. Ναι, πρέπει να τεθεί τέλο όντω και στην απομόνωση. Λείπουν τα τρόφιμα. Εν τω μεταξύ όμω υπάρχει ένα εμπόριο χιλιάδων ε, όπλων. Αν δεν υπήρχε αυτό θα μπορούσαν να μπουν ε, τα τρόφιμα Και αν απαγορευόταν και η εισαγωγή πυράβλων από το Ιράν, θα μπορούσαν να αγοράσουν τρόφιμα. Ε, σταματήσει πια η δημαγωγία. Ε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Μια πολιτική που προβλέπει την ε, χορήγηση πολλών και μεγάλων κονδυλίων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε αυτό το πλαίσιο 7 ε, ετών πολέμου δεν έχει ξαναγίνει. Κανένας από τους συμμάχους μου δεν έπαιξε το ρόλο του. Ή εμάς από το 2008 χρειάστηκε μόνο τέσσερα χρόνια για να προετοιμαστεί από την άποψη την στρατιωτική και έτσι να οργανωθούν και να χρησιμοποιήσουν πολύ σύγχρονους πυράβλους που έχουν πάρει από το Ιράν. Η απειλή λοιπόν δεν είναι η πυρηνική αυτή τη στιγμή, δεν είναι το, το αυτό το πρόβλημα της αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής. το πρόβλημα είναι οι χιλιάδες πύραυλοι οι οποίοι ε, στέλνονται κατά του... Ε, πληθυσμού, του άοπλου πληθυσμού του Ισραήλ και έπειτα η κατάσταση με το Ιράν οι σχέσεις με το Ιράν και με την Αίγυπτο πώς θα συνεχιστούν, πώς θα προχωρήσει η πολιτική που ξεκίνησε ο πρόεδρος της Αιγύπτου σε αυτό το τομέα και έπειτα η πολιτική της Αμάσα στην Λωρίδα της Γάζας. Ορισμένοι συνάδελφοι ακούγοντα ε, όταν μιλούν μου δίνουν την εντύπωση ότι με την ΑΜΑΣ ε, όλα λειτουργούν ειρηνικά στη λωρίδα της Γάζας. Όλα υποτίθεται ότι λειτουργούν φυσιολογικά, ενώ στην πραγματικότητα η Αμάς έχει στρατιωτικούς στόχους και αυτός ο πόλεμος θα περάσει στην ιστορία, γιατί σε μια νέα γεωπολιτική κατάσταση αλλάζει ριζικά η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλαδή την Αμάς με ένα νέο ρόλο, μια νέα σημασία, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν αναλάβει ένα νέο ρόλο με ένα νέο νόημα. Εμείς με την γαθοσύνη ευθύνη μας, παραμένουμε την αφέλειά μας, παραμένουμε και τους κοιτάμε και παριστάνουμε πως δεν έχουμε επιρροή στην κατάσταση. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξέρει η πολιτική μας ομάδα ότι αυτού του είδους η ανακοχή, κατά του πυρός μπορεί να είναι μια ευκαιρία ούτως ώστε να βρεθεί η οριστική λύση μία οριστική λύση. Τέλο πάντων να υπάρξει μία ελπίδα και να μην έχουμε ξανά τη σπίθα που θα φέρει την έκρηξη. Εμείς πρεσβεύουμε ότι η μόνη δυνατότητα, η μόνη λύση είναι το Παλαιστινικό κράτος να υπάρξει. Μόνιμη λύση. Να σταματήσουν επίσης τα εγκλήματα πολέμου, να σταματήσει, το Ισραήλ, να σταματήσει το Ισραήλ να αγνοεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τα όσα λέει ο χάρτη του ΟΗΕ. Τι γίνεται με τις, με συμφωνίες που δεν τις εφαρμόζει όπως τις ε, Τι ε, ε, Τις σχετικές του δεσμεύσεις για να υπάρξει Παλαιστινικό κράτος. Όπως η τελευταία αυτή εισβολή έχουμε ένα σωρό εγκλήματα πολέμου. Έχουμε αυτόν τον αποκλεισμό. Αυτό το εμπάργκο είναι παράνομο κατά το διεθνές δίκαιο. Πρέπει ξεκάθαρα να πάμε προς λύση που περιλαμβάνει συγκρότηση την κράτους. Α, και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα πέρσι είπε ότι είναι υπέρ του να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Παλαιστινικό κράτο με τα σύνορα του 66, το είπε ο πρόεδρο τον είπα. Φυσικά αμέσω <clears throat> διαφώνησε μαζί του Νετανιάχου. Θα πρέπει ομένω να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατόν να καθυστερούμε κι άλλα. Πρέπει να δημιουργηθεί το Παλαιστινικό κράτο. επομένω την 5η 29 του μηνό θα έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία ούτω ώστε να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την συγκρότηση αυτού του κράτους. Δηλαδή αυτό το κράτος αυτό το Παλαιστινιακό να γίνει κράτος που θα μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μην είναι μόνο παρατηρητές. Επίσης ε, έχουμε το 49% των όσων απήντησαν στο Ισραήλ σε ένα γκάλωπ ή δεν ήταν υπέρ της κατάβασης του πυρός. Ήταν σαφώς αντίθεται και στην συγκρότηση του Παλαιστινικού κράτους. Και ο ίδιος ο Μπαράκ, ο Υπουργός, είπε ότι κάνουν μπορούν για να σταματήσει ο αφουγλισμός. Παρ' όλα αυτά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η κοινή γνώμη στο Ισραήλ ζητά ακόμη περισσότερη σκληρότητα. Πάντω, ο αυπλισμό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι μια νοησία αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκόμε. Είναι μια αναγκαιότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ μια επίλυση του Παλαιστινιακού για να μπορέσει το σύνολο τη περιοχή να γνωρίσει την ε, ειρήνη και να σταματήσει ο κινησμός με τον οποίο ακούγονται κάποιες ε, απόψεις ας πούμε τα σχετικά με το Ιράν το οποίο θέλει να έχει πυρνικά για στρατιωτικούς σκοπούς, το δε Ισραήλ επίσης ε, ε, εξοπλίστηκε και έχει τη δυνατότητα να παρέμβει πυρηνικά, να πολεμήσει με πυρηνικά όπλα. Αν έχουμε κάποιο είδου εμπάργκο το οποίο να εμποδίζει το Ισραήλ να εξοπλίζεται με πυρηνικά, αυτό που χρειάζεται να γίνει αποπυρηνικοποίηση τη περιοχή. Αυτά λέει η πολιτική ομάδα και ότι θα πρέπει επομένω από κάθε μετερίζει κανείς να προσπαθεί να βοηθήσει στο να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτο με τα σύνορα όπω είπαμε τα παλιά θα γίνει αυτή η συνεδρίαση των Τούγια, όπου προαναφέραμε και αν μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να είναι παρατηρητές της ε, συνέλευσης, αυτό θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει στη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ πολύ για τον πρώτο αυτό χίρο, αλλά θα πρέπει ίσως να προσπαθήσουμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα για τις στρατηγικές εξελίξεις στο χώρο και όχι μόνο στη Γάζα. Θέλω να τονίσω όμως, γιατί είπατε, Αναγκόμες, κοιτάξτε, εγώ ήμουν στο Στερότ όταν έπεσε μία ρουκέτα αν δείτε λοιπόν πως σε 10 χρόνια έχουν πέσει 10.000 ρουκέτες στα χωριά, δεν μπορούμε να λέμε πως πρέπει να έχουμε κατανόηση μόνο για τους Παλαιστινίους και για τη Χαμάς. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε αντίδραση σε ρακέτες που έπεσαν στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε αυτό. Αυτό ισχύει. Δεν μπορούμε να λέμε πως δεν μπορεί κάποιο να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ανεξαρτήτως το ασκεί λάθο πολιτική, έτσι, με αυτό να συμφωνήσω. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βρίσκουμε μια λύση με βάση τα σύνορα του 67. Α, το ένα οδηγεί στο άλλο. Και οι δύο πρέπει να σταματήσουν τη βία. για να μην επικρατήσουν οι σκληρότερες ε, δυνάμεις. Το να πυροβολούμε δεν το κάνει ο ένας ηθικότερα από τον άλλον και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι σωστό. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για παλαιστινιακά θύματα. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα προς το συμφέρον των απλών ανθρώπων και στις δύο πλευρές. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, πρέπει να δούμε για την κατάσταση του άλλου. Τι πρέπει να κάνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που χρόνια ε, δεν αντιδρά και πέφτουν ρουκέτες. Στην επικράτειά του. αν ξαφνικά προσγειώνονται μια ρουκέτα στη στέγη μου, ε, πόσο να κρατηθεί και μια κυβέρνηση και να μην αντιδράσει. Έτσι. Για να υπερασπίσει και το λαό της. Και στις δύο πλευρές λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να μην υπάρχει βία. Νομίζω αυτό είναι το σωστότερο. και να μην θεωρεί να είναι πιο από τον άλλον εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και τα λέμε και πάλι αύριο.